Ladies and gentlemen, please take a seat. We have now. Καλημέρα σας. Έχουμε ε, ψηφοφορίες σε κάτι εκθέσεις ε, εποσιόδους σημασίας. Σημείο 14. Μαυροβούνιο. Ο Τσάλ Στάνοκ είναι εισηγητής. 15, με συγχωρείτε. Εχθές το βράδυ είχαμε μία συζήτηση ε, ε, με φοβερή οχλαγωγία στις πολιτικές ομάδες να στηρίξουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες υπάρχει αντίρρηση από τους πρασίνους αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής και ξέρετε πού βρισκόμαστε ωραία οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με την παράγραφο 1 τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές για το 10. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν προφανές, μάλλον απορρίφθηκε, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. «41 υπέρ, 20 όχι». 16 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 19 αποσύρεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά Ατυχώς για σας απαντάει ο πρόεδρος σε ένα σχόλιο χωρίς μικρόφωνο. Λίγη ψηφοφορία. όντως ε, ατυχές για σας 34 υπέρ 33 κατά 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 με μία προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κα, κατά αποχές εγκρίνεται πρώτη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τριάντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Διότι πολλοί νομίζω δεν ψήφισαν, άρα παίζεται. 52, τροπολογία 52. Λίγη τροπολογία, η ψηφοφορία για την 52 εγκρίθηκε με 38 υπέρ 28 κατά. 53. 53 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 54 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 νομίζω είναι η επόμενη. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο underlines έως charter ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιατί τότε κάναμε και τα δύο τμήματα τέλος πάντων. 60. Με την ε, προφορική τροπολογία του κυρίου Βάγκελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη ηλεκτρονικός έλεγχος λίγη Απερίφθη 29 υπέρ 35 κατά. 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 63 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 64 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 65 υπέρ κατά εγκρίθηκε 66 υπέρ κατά εγκρίθηκε 67 υπέρ κατά εγκρίθηκε 68 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίθηκε με την ίδια ε, πλειοψηφία όπως και πριν. 69 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 70 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 71 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 72 υπέρ κατά απερίφθη 73 υπέρ κατά εγκρίθηκε 74 υπέρ κατά εγκρίθηκε 75 υπέρ κατά απερίφθη 22 ε, Δύο, δύο με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Είναι νωρίς το πρωί και ε, διπλοβλέπω φαίνεται. Απερίφθη όμως. Ε, τρία και τέσσερα υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Πέντε υπέρ κατά απερίφθη 6 κατά απερίφθη 7 υπέρ ηλεκτρον... ηλεκτρονικός έλεγχος για το... την τροπολογία 6 λίγη Λοιπόν, ενεκρίθη. 7 υπέρ, κατά. Και πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη ψηφοφορία. Απερι... Ε, 40 υπέρ, 26 κατά υπάρχει μία μυστική πλειοψηφία σιωπηλή η οποία δεν εκφράζεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Ποιος είναι υπέρ της ε, τροπολογίας 1. Υπέρ. Κατά. Ενεκρίθη. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. ενεκρίθη 60 υπέρ 2 κατά και καμία αποχή. Συγχαίρω τον Τσάρλς σαν εισηγητή. Λοιπόν, προχωρούμε. Πάμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η είναι η κυρία Ντόρις Πακ. Έχεις να πεις τίποτα. Θα σας παρακαλούσα να είστε προσεκτικός στην ψηφοφορία και ή δυνατόν να ακολουθήσετε εμένα. Υπάρχουν δύο τροπολογίες που θεωρώ ότι βλάπτουν περισσότερο παρά εξυπηρετούν. Κυρία Πακ, ποιος τολμάει καν να είναι αντίθετος με τις προτάσεις σας, αν είναι δυνατόν. Προσωπικά ουδέποτε το επιχείρησα. So. Λοιπόν, συμβαστική παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ Κατά, κατά εγκρίνεται. Εποχές. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Τι θέλετε, έλεγχο για το πρώτο τμήμα, μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 42 υπέρ, 24 κατά. Το δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην 24 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές 28 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική 5 λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 45 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 50 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 54. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου ε, εποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αυτό θέλει έλεγχο Άρχιψη, ψηφοφορία πέρασε 29 υπέρ 38 κατά απορρίπτεται 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 57 υπέρ κατά απορρίπτεται 58 υπέρ κατά απορρίπτεται 59 υπέρ κατά εγκρίνεται η 60 υπέρ κατά εγκρίνεται υπέρ 61 συγγνώμη κατά Εγκρίνεται. 6. Η συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Συμβιβαστική. Κατά. Εγκρίνεται. Η 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Ε, η κυρία Κορνέλησεν. Ναι. Θα παρακαλούσα να κάνω μια προφορική για τη συμβαστική υπαριθμών 8. Να αφαιρεθούν οι λέξεις ανησυχεί για τον εξτρεμισμό μέχρι να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Καλεί τις αρχές χώρας να καταπολεμήσουν τον εξτρεμισμό ε, τη μυσαλλοδοξία σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα για να ε, ληφθούν ε, εξεμιστικές και ακραίες απειλές κάθε είδους παντού στην επικράτεια των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ντόρις. Εχθές κάναμε συμβιβασμό, εγώ παραμένω στο συμβιβασμό, για, συμβιβασμό γιατί είναι αντικειμενικός, δεν υπερβάλλουμε. Πριν έρθει το τσουνάμι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην μας κατακλείσει. Μάλιστα. Ψηφίζουμε λοιπόν το συμβιβασμό. 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ορίστε. Όχι, δηλαδή απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 75 υπέρ κατά εγκρίνεται 76 έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ Ich entschuldige mich ausdrücklich für Ζητώ συγγνώμη για τον αντιπρόεδρό μου που είπε ότι σεξου... ε, καλωσορίζει τη σεξουαλική βία η τροπολογία. Αστιάκη. Υπέρ του πρώτου τμήματο παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Και μετά το επόμενο υπέρ κατά δεν είναι σαφές όμως. Η ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται ισοψηφία. 77 και πάλι κατά τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλωσορίζει τα βασανιστήρια, λέει ο πρόεδρος τώρα. Τώρα κατάλαβα γιατί αποφάσισε η ομάδα μου να καταψηφίσει το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Και αυτό χρειάζεται έλεγχο νομίζω. Αλλά μάλλον να εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κατά. Das τη ist Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 79. Όχι, έχει αποσυρθεί. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δηλαδή απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 85 υπέρ. Κατά. Η συμμετοχή φθήνει όλο και περισσότερο. Παρακαλώ να ψηφίζετε. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 84. Της 85. 33 υπέρ, 34 κατά απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά εγκρίνεται η 91 υπέρ κατά απορρίπτεται η 92 υπέρ κατά απορρίπτεται Απορρίπτεται. Πού είμαστε τώρα. 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά απορρίπτεται 90 dafür 99 υπέρ κατά εγκρίνεται 100 υπέρ κατά απορρίπτεται έλεγχο θέλετε άρχεται η ψηφοφορία για την αριθμό είναι 100 100 δεν είπαμε ναι. 32 υπέρ, 34 ε, κατά, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά. Θέλει έλεγχο και αυτό. Μάλλον να έχει απορριφθεί, αλλά δεν ήταν σαφές. η ψηφοφορία. Λίγη. 33 υπέρ, 37 κατά απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. 31 υπέρ, 35 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110, όχι, καλύπτεται αυτή. 111, υπέρ. Κυρία Μποσκούρτ θέλει το λόγο. Συντάκτρια της τροπολογίας. Θα ήθελα να προτείνω μια προφορική ε, τροπολογία για το τελευταίο τμήμα της 111, γιατί με ενημέρωσαν από την Κροατία ότι το τελευταίο, ε, αυτό που αφορά τη γέφυρα, έχουν σταματήσει ε, οι διαδικασίες ανέγερσης. Ε, η Κροατία έχει σχέδια ανέργησης για τη γέφυρα του Πέλιασατ, στα οποία αντιτίθεται η Βοσνία Ζεγοβίνη. Ε, θα μπορούσαν να βλάψω τη μελλοντική ανάπτυξη, λέει του Βοσνιακού Λιμέν η Πρόεδρος. Αν δώσει τα λεφτά η κυρία Μποσκούρτ στη Βοσνία, και στη, τα λεφτά θα, τα, θα τη φτιάξει τη γέφυρα και στην Κροατία. Η Κροατία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει καμιά σχέση με τη Βοσνία, έχει σχέση με τον προπολογισμό. Ε, λοιπόν, ας μην ε, ζητάμε παράλογα πράγματα, διαφωνώ με αυτή την τροπολογία. Είναι οικονομικό το ζήτημα. Ναι, μπορούμε να ψηφίσουμε, θέλετε, την πρόταση για την 111. Για την 111 δεν είπατε την προφορική τροπολογία. Ε, όπως πρότεινε προφορικά η κυρία Μποσκούρτ. Μα δεν γίνεται όταν κάνει κάποιος μια τροπολογία ε, να, να αλλάζει με προφορική τροπολογία την ίδια της τροπολογία. Η κυρία Μποσκούρτη την έχει κάνει την 111, προτείνει μια προφορική αλλαγή της τώρα. Έχει δίκιο η Ντόρις. Ε, όταν διαφωνεί κάποιος Μα κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρο, ε, δικέ σου τροπολογίε δεν μπορεί να τι αλλάζει. Προφορικά. Η ε, κυρία Πακ χωρί μικρόφωνο. Είναι ένα καινούριο σημείο. Κατηγορεί μια γειτονική χώρα ε, που δεν κατασκευάζει μια γέφυρα. Ε, δεν μπορεί η χώρα αυτή, δεν δύνατη γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς κανονίζουμε τον προϋπολογισμό της Κροατίας δεν έχει καμία σχέση με την έκθεση για τη Βοσνία. Απλώς περνάει και από τη Βοσνιακή επικράτεια η γέφυρα. Ξέρετε όλοι ποια είναι η οικονομική κατάσταση όλων και της Κροατίας. Τώρα θα πρέπει να την αναγκάσουμε να φτιάξει αυτή τη γέφυρα που δεν έχει τα λεφτά. Ψηφίζουμε την 111 με την αρχική μορφή, λέγει ο Πρόεδρος. Και παρακαλείται η κυρία Μποσκούρτ να καταθέσει την τροπολογία της στην Ολομέλεια. 111 ψήφι υπέρ. Υπέρ της αρχικής μορφής. Ή ε, κατά είμαστε, λέει η κυρία Πακ ε, που τα έχει μπλέξει. Ε, 111 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Yeah. Lächerlich. Kommt 33 υπέρ, 35 κατά απορρίπτεται. Γέφυρα Γιόκ. 112. Της κυρίας Λούνατσεκ. Μάλλον το λόγο έχει η κυρία Λούνατσεκ. Εγώ δεν κατάλαβα τι ψηφίσαμε τώρα. Νόμιζα ότι ψηφίσαμε την αρχική τροπολογία. Α, εντάξει, τότε καλά ψήφισα. Την αρχική τροπολογία 111 ψηφίσαμε. 112 υπέρ κατά απορρίπτεται η προφορική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά απορρίπτεται υπέρ τις 5 κατά εγκρίνεται η 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 9 με την προφορική υπαριθμό 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 11 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 13. Σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το τρίτο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 15 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Γιατί 15. Πέρας. 32 zu 38 abgelehnt. 32 υπέρ, 38 κατά απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 1 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 2 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ποιο είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρο τώρα. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. Εγκρίνεται 58 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 9 αποχές. Συγχαρητήρια, Ντόρις. Can you share for two minutes? Peter. Ε, λοιπόν, συνεχίζουμε. Να περάσουμε στη Σερβία. Ψήφισμα για τη Σερβία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Πρόεδρε. Κυρία Κατσίν, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, πριν ξεκινήσουμε. Να προτείνω μια μικρή αλλαγή στην, αλλαγή, στην τροπολογία 153. Θα ήθελα το Μακεδονία να αντικατασταθεί από Φύρομ. Μία επισήμανση των Ελλήνων φίλων και είναι αποδεκτή. Και να εξηγήσω και την θέση μου για τις τροπολογίες 113 και 14. Για την 113 έχουμε να κάνουμε τη βλάχη και μειονότητα και μετά με την αλβανική στην 114. Βουλγαρική. Βουλγαρική. Εδώ λοιπόν θα απευθύνω επιστολή στις σερβικές αρχές για να εξηγήσουμε ότι θα παρέχεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των μειονοτήτων σε όλη τη Σερβία, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής. Αυτό που θέλουμε είναι οι βλάχοι να έχουν την ίδια προστασία όπως και η βουλγαρική μειονότητα. Αυτό θα, η επιστολή θα αποσταλεί την επόμενη εβδομάδα. Οπότε ελπίζουμε ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων θα βελτιώσει την παρούσα κατάσταση στην κεντρική Σερβία. Πρόεδρος, Νομίζω όλοι κατάλαβαν τη θέση σα σχετικά. Είναι να περάσουμε στην προφορία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Για την 153. Δεν κάνουμε συζήτηση. Μα συγγνώμη, πρότεινε προφορική τροπολογία. Okay. Εντάξει. Compromise 1. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23 Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Compromise number. Compromise 2. Who Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εκτός μικροφώνου. 29. Υπέρ. Κατά. εγκρίνατε. 30 υπέρ. 30 υπέρ. Κατά. Νομίζω να κάνουμε έναν έλεγχο καλύτερα. 30. Για την 30. The boat is closed. Πέρας. Απορρίπτεται 34 προς 30. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40. Συμβαστική 4 μάλλον. Πρόεδρε, μια προφορική τροπολογία στο τέλος της συμβαστικής 4, τελευταία πρόταση που λέει καλώς αρίζει τους φραγμούς από την πλευρά της σερβικής, από τη σερβική πλευρά, νομίζω η σερβική πλευρά των διοικητικών συνόρων θα πρέπει να αλλάξει στο Σερβία. Απορρίπτεται. Compromise stands. In Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51. Με δύο προφορικές τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. 59. Σέπφλιν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Με τις διαγραφές όπου δεν θέλουμε να δυναμώσουμε τη στρατηγική, υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 78 σε δύο τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ Τη συμβαστική 8. Κατά. Εγκρίνεται. Εβδομήντα 73 τώρα. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμμεπαστική 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σωστά. Έλεγχος. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 27 προς 41. 114 υπέρ κατά απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Έλεγχος, μάλιστα. Σχεδόν έληξε ψηφοφορία. Τώρα έληξε πραγματικά. 28 προς 37 απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμμεπαστική 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 126, 126 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. 13. συμβαστικά 13 ΕΠΕΡ Κατά. Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 135. Θα έπρεπε να ψηφίζουμε μέχρι 135 όσο έχει. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 137. Καταπίπτει. 138 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. το ΕΛΚ. Αν δεν ψήφισε το ΕΛΚ, θα έχει εγκριθεί. Εγκρίθηκε. Καλά, ας ελέγξουμε. Υπέρ. Okay, course. Okay. Now it's stopped. Πέρας. Μετά από εντατικέ συζητήσει στο ΕΛΚ, η ευρεία πλειοψηφία του 55 προ 10 οδηγεί στην έγκριση. 141 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 140. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. 142. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 143. Κατά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα. 152. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Uh, Κυρία Μπρέντνερ, εδώ έγινε προφορική τροπολογία από τον κύριο Κατσίν για την ε, προσθήκη του, της Φύρομ. Πράγμα που απορρίπτω. Μακεδονία αναφέρεται στο κείμενο. Να μείνει ως έχει. Ναι, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούμε την επίσημη ορολογία στα ψηφίσματά μας. No, but we can say that we are Κοιτάξτε, μπορούμε να καταψηφίσουμε, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σωστή ορολογία. Συγγνώμη κύριε Μπροκ. Μα το πολιτικό ζήτημα στην περιοχή είναι ακριβώς το, η ονομασία. Δεν είναι θέμα τεχνικό, τεχνικής επιλογής. 153. Ψηφίζουμε την 153 υπέρ. Ως έχει, ως έχει. Κατά. Εγκρίνεται. 54. But this it is part which is already decided to compromise now. Στη συμβαστική 9, το τμήμα που ήδη έχει υπερψηφιστεί, θα διαγραφεί από εδώ. 154 υπέρ, κατά Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. It was clear. Otherwise we should must vote. Αν δεν είναι σαφές να ξαναψηφίσουμε. Για μένα ήταν σαφέστατο ότι απορρίπτεται. little bit faster. Λίγο γρηγορότερα. We take, we take the Μόνο ένας να μετράει. Έτσι λέει και ο Πούτιν. Δεν έχει σημασία ποιος ψηφίζει, ποιος μετράει. Έχει σημασία. Can I close the Yeah, it's closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 προς 40. 155. Υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται με την ίδια αναλογία. 157. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 158. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Μοιάζει να απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 προς 41. Συμβαστική 15 υπέρ. Όχι, 159 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 163. Καταπίπτει. 166 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 προς 39. Συμβαστική 16. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 176. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 177. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 5 υπέρ, Κατά. Πέντε υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε από τους μισούς από τους ψηφίσαντες, άρα απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Δεν ψήφισαν ούτε μισή. Εντάξει, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όσοι τουλάχιστον είναι υπέρας, ψηφίσουν. Καλό θα ήταν να την περάσετε. Πέρας. Θα σας παρακαλούσα πραγματικά να ψηφίσετε. 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική εκδοχή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 62 προς 4 και με 5 αποχές. Εάν ο κύριος Τάρνοκ μας προσφέρει τουρκικό καφέ, ευχαρίστως να κάνουμε διάλειμμα. I have Λοιπόν, ε, ορισμένες ε, τροπολογίες έχουν αποσύρθει από την κυρία Μπόσκουρτ και από την κυρία Σόμερ και οι συνάδελφοι είναι ευτυχείς, δηλαδή θα μειωθεί η ψηφοφορία. Η κυρία Όμεν Ρόιτερ έχει κάτι να μας πει. Ναι, Kompromiss 1 dafür. Dagegen Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 69. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά απορρίπτεται 71 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά απορρίπτεται 70 ε, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 77 υπέρ κατά πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος 77 ο κύριος Λάμπσδορφ Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία σάφια ε, στον κατάλογο ψηφοφορίας. Η Χάουιτ απορρίπτεται, αλλά ε, εάν ισχύσει η 73, αλλά η 73 ε, καταρρίπτεται εάν υπερψηφιστεί η συμβαστική 2. Άρα πρέπει και οι δύο αυτές να μην προχωρήσουν. Κυρία Ομαν Ρόιτερ. Έχει δίκιο ο κύριος Λάμστον. Χθε έγινε ένα σχόλιο όμως από τον κύριο Χάουιτ και για το λόγο αυτό το βάλαμε σε ψηφοφορία γιατί υπάρχουν κάποιες λέξεις που διαφέρουν και θελήσαμε να μην γίνει συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο έφτασε στην ψηφοφορία. Εάν συμφωνεί όμως... Για μένα εμπίπτει, καλύπτεται από το συμβιβασμό, αλλά εξαρτάται του τον κύριο Χάουιτ το κανόνισα με τον κύριο Μπιόλς, ο οποίος ασθενεί και του εύχομαι περαστικά, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, αλλά ο κύριος Χάου ε, δεν θέλησε να το σεβαστεί. Εάν ε, τώρα το δέχεται, ε, εντάξει. Welche reden wir denn jetzt? 73 oder 77? Ja, Sie reden aber über Obiols. Ja, Obiols war der Schattenberichterstatter. Hat gesagt, es war abgedeckt. Aber Howitt okay. nicht. Then, uh, äh, Mr. Howitt. Λοιπόν, κύριε Χάουιτ, Εάν η πρόθεση είναι να υπάρξει διακριτική ευχέρεια δεν επιτεύχθη ο στόχος. Εγώ είπα ότι θα έπρεπε να διευρύνουμε την ενέργεια που δεν περιλαμβάνεται στην συμβιβαστική 2 οπότε ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον εσωτερικό κανονισμό. Θα πρέπει να ψηφιστεί. Λοιπόν, ο εισηγητής θεωρεί ότι καλύπτεται, ο κύριος Χόουιτ όμως θεωρεί ότι δεν καλύπτεται, οπότε η ψηφοφορία θα αποφασίσει. 77. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απερίφθη. Να κάνουμε όμως ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 77 του κυρίου Χάουιτ. Ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη. 26 υπέρ, 37 κατά. 84 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ενενήντα. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους, κατά, Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 91. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στην 98. και πάλι σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Απορρίπτεται. Και πάλι με ε, ε, κακή συμμετοχή των συνεργατών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία 101 ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. 22 υπέρ, 43 κατά, απερίφθη. Νομίζω ότι υπήρχε κάποια μικρή διαφορά. Να ξαναελέγξουμε. 103 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι, Απερίφθη 29 υπέρ 34 κατά. Συμβιβαστική 5. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ κατά απορρίπτεται 6, 106 υπέρ κατά εγκρίνεται δεκαοχτώ σε δύο τμήματα ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 118 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος νομίζω ότι απερίφθη αλλά ας το ελέγξουμε διότι μετά θα έρθει ένας πρωθυπουργός οπότε πρέπει να τελειώσουν τις ψηφοφορίες έχοντας καλά ελέγξει τι κάναμε απερίφθη Ερχόμαστε στη συμβιβαστική 7. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Στην 123 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά απορρίπτεται 137 υπέρ κατά εγκρίνεται 'Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να συμμετέχετε στην ψηφοφορία. 40 έως 50% των μελών της Επιτροπής ως επιτοπλίστων δεν ψηφίζουν. Ακόμη και τώρα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία ο Τσάλς Τένοκ δίκιο είχε έπρεπε να κάνουμε διάλειμμα για καφέ. Έληξε. Εγκρίθηκε 38 υπέρ 25 κατά. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά Εκατόν σαράντα ηλεκτρονικός έλεγχος. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος είναι εκατόν σαράντα. Έληξε. Ενεκρίθη 37 υπέρ 29 κατά 145 που είναι ενδιαφέρον από πλευράς ηλικία. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά απορρίπτεται Νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο διότι ορισμένα μέλη δεν συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. 147. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. 56 υπέρ, 10 κατά. Ήταν λοιπόν καταφανές. Αλλά επαναλαμβάνω μία ακόμη φορά σας παρακαλώ να συμμετέχετε στις ψηφοφορίες ιδίως όσοι θέλουν να επικροτήσουν διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. 149 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Απορρίπτεται. Για το δεύτερο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 152 και 161 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 153 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ε, Ρία, κοίταξε τι, τι, λες αν, είναι, αν είσαι υπέρ ή κατά, αλλά το έλκος επτοπλίστων δεν ψηφίζει. Το 153 υπέρ. Λίγοι. 39 υπέρ 27 κατά. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 170. Υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. 171. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 176 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος.

με αυτή την τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 397 σαν προσθήκη στην τροπολογία 13 υπέρ κατά απορρίπτεται 189 σε τρία τμήματα για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται τώρα ερχόμαστε στη 14η συμβιβαστική ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 211 υπέρ κατά απερίφθη 213 υπέρ κατά απορρίπτεται 215 υπέρ κατά εγκρίνεται 216 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 217 υπέρ σε τρία τμήματα ένα υπέρ κατά εγκρι... απερίφθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται τρίτο υπέρ κατά Απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 222 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 223 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 224 υπέρ κατά απορρίφθηκε συμβιβαστική 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 228 υπέρ κατά απορρίπτεται 235 υπέρ κατά απορρίπτεται 237 υπέρ κατά απορρίπτεται 238 υπέρ κατά απορρίπτεται 240 σε δύο τμήματα υπέρ κατά απορρίπτεται Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 248 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 250 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 250. Λίγοι. 10 υπέρ, 53 κατά. Συμβιβασμός 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. ...252 υπέρ, κατά, απορρίπτεται με τη συμμετοχή 10% των συμμετεχόντων απερίφθη. Απερίφθη 252. Ε, ε, ε, η καταπίπτη εάν ε, εγκρινόταν η συμβιβαστική 19 που δεν, που δεν ε, εγκρίθηκε και η 252 απερίφθη, 253 τώρα υπέρ, κατά, απερίφθη. 254 υπέρ, κατά, Απερίφθη. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 264. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 200, ε, συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 271 αποσύρεται, 272 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 274 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 277 υπέρ, κατά απορρίπτεται 281 υπέρ κατά εγκρίνεται 352 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 282 υπέρ κατά απορρίπτεται 283 υπέρ κατά Εγκρι... απορρίφθηκε 284 υπέρ κατά απορρίφθηκε 285 υπέρ κατά απορρίφθηκε 286 υπέρ κατά απορρίπτεται 287 υπέρ κατά απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος έληξε ενεκρίθη με 35 υπέρ και 30 κατά. 288 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 289 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 290 υπέρ κατά απορρίπτεται 291 πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ Λοιπόν, 292. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, υποθέτω, του 291. Λίγοι. Απερίφθη. 292 υπέρ κατά απερίφθη 293 υπέρ κατά απερίφθη 294 υπέρ κατά εγκρίνεται 295 υπέρ κατά εγκρίνεται 298 υπέρ κατά εγκρίνεται 296 υπέρ κατά απορρίπτεται 297 υπέρ κατά απορρίπτεται 299 υπέρ κατά υπέρ 299 κατά απερίφθη 300 υπέρ κατά απερίφθη κύριε Λάμπστορφ ο πρόεδρος παρακαλώ μπορεί να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο που είναι πιο κοντά στο κάθισμά του γιατί πολλές φορές δεν τον καταλαβαίνουμε. Ε, ίσως ο κύριος Λάμπστορ νομίζω ότι αυτός θα έπρεπε να ηγείται της ομάδος. Έτσι είναι όλοι τους οι φιλελεύθεροι. 303 ε, υπέρ, κατά, καταπίπτει. 305 υπέρ κατά απερίφθη. 306 υπέρ κατά απερίφθη. 308 υπέρ κατά απερίφθη. 309 υπέρ Λίγοι από τους 71 παριστάμενοι μόνο 57 ψήφισαν και απερίφθη με 15 υπέρ και 42 κατά. Η 309 υπέρ κατά. Απερίφθη. 310-311 υπέρ κατά. Απερίφθη. 312 υπέρ κατά απερίφθη 315 υπέρ κατά απερίφθη 316 υπέρ Μα έχουμε 316, γιατί 317 το 316 απεσύρθη, 317 υπέρ κατά απερίφθη. 318 υπέρ κατά απερίφθη 319 και 326 υπέρ κατά απερίφθη Τι έγινε, υπάρχουν δύο ίδια άτομα τα οποία υπέβαλαν δύο φορές τις ίδιες τροπολογίες. Μπας και μία χαρανότα στο δρόμο. 320. Ε, Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 321. Υπέρ. Έχει πάλι αποσυρθεί. Θα έπρεπε να μας το λένε. 322. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 323. Η 322 απερίφθη. 323 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχέσε. απορρίπτεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 329 υπέρ. Κατά. Ε, Απορρίπτεται. 331 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 334 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 335 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 336 υπέρ κατά απορρίπτεται 337 υπέρ κατά απορρίπτεται 338 υπέρ κατά απορρίπτεται 339 υπέρ κατά απορρίπτεται 340 υπέρ κατά απορρίπτεται 342, 43 και 44. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 345 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 347 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 348 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 349 υπέρ κατά απορρίπτεται 350 υπέρ κατά απορρίπτεται 351 υπέρ κατά απορρίπτεται 354 υπέρ κατά εγκρίνεται 355 υπέρ κατά απορρίπτεται 357 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 359, 60, 61 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 364 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 366 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 367 υπέρ κατά απορρίπτεται 371 υπέρ κατά απερίφθη υπέρ κατά απερίφθη 368-69 υπέρ κατά απερίφθη 370 υπέρ κατά απερίφθη 372 υπέρ κατά απερίφθη κύριε Λάμστορφ σχετικά την 373 έχουμε μία προφορική τροπολογία διότι ίσως μάθατε ότι το, το συνταγματικό ο δικαστήριο της Γαλλίας απέριψε ε, την ε, γενοκτονία των Αρμενίων ως ε, εγκληματική πράξη οπότε θα θέλαμε να υπάρξει μία προφορική τροπολογία η οποία προβλέπει άνοιγμα των συνόρων και με στόχο να μπορέσει να μην ψηφίσει κανείς Έχει περιληφθεί η προφορική τροφολογία. Ποιος έχει τη σωστή ε, προφορική τροπολογία 373, ποιος είναι κατά. Απέρευτη. Πάμε στη 376. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 374, υπέρ κατά εγκρίνεται 375 υπέρ κατά απορρίπτεται 377 υπέρ κατά απορρίπτεται 378 υπέρ κατά 378 υπέρ, κατά απορρίπτεται 380 υπέρ κατά απορρίπτεται 381-384 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 382 υπέρ κατά απορρίπτεται 383 υπέρ κατά απορρίπτεται 385 υπέρ κατά απορρίπτεται 76 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 74 υπέρ κατά απορρίπτεται 386 υπέρ κατά απορρίπτεται 388 υπέρ κατά απορρίπτεται 390 υπέρ κατά απορρίπτεται 391 υπέρ κατά απορρίπτεται 393 υπέρ κατά απορρίπτεται υπέρ κατά το 396 απορρίπτεται 398 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 23 υπέρ κατά εγκρίνεται έτσι ερχόμαστε στην 404 υπέρ κατά απορρίπτεται 405 καταπίπτει και συνέχεια 408 υπέρ κατά απορρίπτεται 411 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 418 υπέρ κατά απορρίπτεται 419 υπέρ κατά εγκρίνεται 421 υπέρ κατά απορρίπτεται 421 ηλεκτρονικός έλεγχος Λίγοι. Ενεκρίθη 37 υπέρ 26 κατά και μία αποχή. Οπότε πάμε στο 422 η οποία θα συγχωνευτεί με την 421 για να μην υπάρξει συγχώνευση, ε, να μην υπάρξει σύγχυση, 422. Απερίφθη. 423 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ενεκρίθη, διότι αυτή τη φορά οι φιλελεύθεροι επεκρότησαν, υπερψήφισαν. Λοιπόν, ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 423. λίγη I have not a feeling that everyone follows this line. 424 dafür. 424 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 425 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 426 υπέρ κατά απορρίπτεται 427 υπέρ κατά εγκρίνεται 428 υπέρ κατά απορρίπτεται 429 υπέρ κατά απορρίπτεται 430 υπέρ κατά απορρίπτεται 431 υπέρ κατά απορρίπτεται 432 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 24 υπέρ κατά εγκρίνεται και ερχόμαστε στην 433 υπέρ κατά απορρίπτεται 434 υπέρ κατά απορρίπτεται 438 υπέρ κατά απορρίπτεται 440 υπέρ κατά απορρίπτεται 442 υπέρ κατά απορρίπτεται 443 υπέρ κατά απορρίπτεται 445 υπέρ κατά απορρίπτεται αλλά χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν ήταν σαφές εδώ. Για την 445. Λίγοι. 12 υπέρ 50 ε, κατά. 446 υπέρ κατά απορρίπτεται 448 υπέρ κατά απορρίπτεται 449 υπέρ κατά εγκρίνεται 450 υπέρ κατά εγκρίνεται 451 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη με 29 υπέρ και 30 κατά. 452 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 455 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 458 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι για το πρώτο τμήμα του συνολικού συστήματος, ποιος είναι για το δεύτερο. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 459 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 460 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 461 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά απορρίπτεται 8 υπέρ κατά απορρίπτεται 9 και 10 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι το 9 και το 10 δεν είναι ταυτόσημα γιατί και τα δύο προσθέτουν ε, στο τέλος with the aim of accession αλλά το 9 κρατά όλη την ε, παράγραφο δηλαδή ε, για open-ended process. Δεν είναι δηλαδή ταυτόσημες αυτές οι δύο τροπολογίες. Οπότε πρέπει να τις ψηφίσουμε χωριστά. Ξεκινάμε και ψηφίζουμε την εννέα. Ποιος είναι υπέρ της εννέα. Κατά. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Επίσης απερίφθη. 11. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 12. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Δεκατρία Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 14 υπέρ κατά απερίφθη 15 υπέρ κατά απερίφθη 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά απορρίπτεται 19 και 20 υπέρ κατά απορρίπτεται 21 υπέρ κατά απορρίπτεται 22 σε 2 τμήματα ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά απορρίφθηκε για το δεύτερο τμήμα υπέρ ε, κατά επίσης απερίφθη 23 υπέρ κατά απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 24, ο κύριος Λάμπστορφ. Σχετικά με την 24 υπάρχει μία προφορική τροπολογία η οποία μου φαίνεται παράλογη γιατί λέγεται ότι αν καλυφθούν οι προϋποθέσεις στα πλαίσια της διαδικασίας θα ανοίγουν κεφάλαια αλλά ε, εάν θίγεται η κυριαρχία κρατών μελών για κάθε κεφάλαιο δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται ότι πλήγεται η κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν θα κάνουμε συζήτηση επί του περιεχομένου περιεχομένου ε, εάν η, λογική της ψηφοφορίας είναι ότι αποκλεί τα παράλογα. Αλλά εγώ είμαι ενάντιος και η ομάδα μου εις ε, αυτήν την προφορική τροπολογία και ζητούμε να μην γίνει αποδεκτή προφορική τροπολογία. Ωραία. Οπότε η 24 θα ψηφιστεί χωρίς προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 25 υπέρ. Καλύπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28, 29, 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 32 υπέρ κατά απορρίπτεται η 35 απεσύρση, 36 υπέρ κατά απορρίπτεται 37 υπέρ κατά απορρίπτεται 39-40 υπέρ κατά απορρίπτεται 38 υπέρ κατά απορρίπτεται 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 υπέρ κατά απορρίπτεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 υπέρ κατά απορρίπτεται 46 υπέρ κατά απορρίπτεται ε, συμβιβαστική 27 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 28 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 29 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 64 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά. Εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ένα, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερη τροπολογία, υπέρ. κατά εγκρίνεται. Τρία, υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφο, τελική ψηφοφορία. Ja, Die Abstimmung ist geschlossen. Λίγη ψηφοφορία. Η έκθεση έγινε αποδεκτή με 54 ψήφους υπέρ 7 κατά. Ε, συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα να με ακούσετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο το προσωπικό, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά ε, και αυτή τη φορά όλες ε, τους συναδέλφους ε, της πολιτικής ομάδας, της γραμματείας της Επιτροπής, τους προσωπικούς μου συνεργάτες και βοηθούς. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι για τον κύριο Μπιόλς, καλά λόγια, ο οποίος ασθενεί σήμερα, και όλους τους κοιόδες συγητές. Είχαμε πάρα πολύ καλή ε, συνεργασία και σας ευχαριστώ πολύ. Äh, Οι επόμενες ψηφορίες την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ακόμα τρία τέταρτα. Δεν γίνεται. Είναι γνωμοδότηση ε, για το PNR. Αυτή πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ των τροπολογιών. Τώρα ψηφίζουμε για το PNR. Δεν παίρνουμε ε, το λόγο. Ουγγουράν. Ένα έως τέσσερα τροπολογίες. Κατά. Απορρίπτεται. Το σύνολο. Υπέρ της γνωμοδότησης ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τσεκ φωνάζει η κυρία και εκτός μικροφώνου. Υπέρ της γνωμοδότησης ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είμαστε στην τελική ψηφοφορία της ε, γνωμοδότησης Ουγγουράνου, υπέρ. Στην τελική ψηφοφορία. Πού? Bitte stimmen Sie ab noch. Es sind erst 43 ab. Παρακαλώ ψηφίστε, δεν ψηφίζετε. Πέρας ψηφοφορίας. Επανάληψη. Ψηφίζουμε ε, τη γνωμοδότηση ε, Ουγγουρεάνου, ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση για το PNR. Τις τροπολογίες τις ψηφίσαμε. Ένα έως και τέσσερα. Καταψηφίστηκαν. Ναι, αλλά θέλουν ηλεκτρονικό έλεγχο οι πράσινοι. Όποιος δεν ψηφίζει και χάνει την ψηφοφορία θέλει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Να συμμετέχετε στις κανονικές ψηφοφορίες. Τελευταία φορά το κάνω. Την άλλη φορά όχι. Όποιος δεν ψηφίζει. Λοιπόν, τροπολογίες 1 έως 4. Κατά. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης, επαναλαμβάνω. Now the vote is closed. Πέρασε. 26 υπέρ, 12 ε, κατά, 13 αποχές. Ο κύριος Λάμστορφ είχαμε κανονικό χρονοδιάγραμμα ε, για ε, να ψηφίσουμε ε, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Αύριο υπάρχει συνεδρίαση. Ήθελε η Γραμματεία να ψηφιστεί για να έχουμε σαφή εντολή για να μπορέσουμε αύριο στην ομάδα εργασίας να έχουμε εντολή. Για την Τουρκία είχαμε χρόνο. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η πίεση. Έχουμε πολλές συμβαστικέ προτάσεις. Μπορεί να ψηφιστεί πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα ε, του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μπορούσατε να το είχατε πει ε, προηγουμένω. Ε, ψηφίσαμε σήμερα το πρωί πάνω από χίλιε τροπολογίε. Ήταν πάρα πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Και έχουμε τον Σέιχη πρώτων πυλών. Τι να τον αφήσουμε να περιμένει. Μπορεί εγώ να είμαι ανοργάνωτος, αλλά τι να κάνω, έτσι είμαι. Κύριε Λάμσταρ, να, λέτε στην αρχή της ε, ε, ψηφοφορίας να ψηφίσουμε πρώτα το θέμα σας και όχι τελευταίο, για να βοηθάμε ένα τον άλλο. Την Τουρκία έπρεπε να την είχαμε ψηφίσει την άλλη εβδομάδα. Αν προλάβουμε στις 12, μπορούμε να προσπαθήσουμε να το ψηφίσουμε σε περίπτωση που τελειώσουμε. Αλλά τώρα θα δεχτούμε τον Πρωθυπουργό του Κατάρ. Παρακαλώ. Ή δυνατό μετά τη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό κατά τις 12 θα κάνουμε και άλλη ψηφοφορία για το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Κυρίε και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Μετά από δύο ώρες εντατικών ψηφοφοριών, είμαστε λίγο κουρασμένοι. Αλεξάνδρ, κάθισε σε παρακαλώ. Θα δούμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία αργότερα. Θέλω να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, που είναι και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας του. Σας ευχαριστούμε που έχετε έρθει σήμερα εδώ. Ξέρουμε ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Λόγω και των αλλαγών στην Βόρεια Αφρική, τη Συρία, Και έτσι θεωρώ ότι η αυτοξοχότητά σας μπορεί να προεδρεύει και στην, στο σύνδεσμο των αραβικών κρατών και βεβαίως παρεμπρεθήκατε και στην 66η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε την απόψη σας αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω. Θα σας δώσω το λόγο, Πρωθυπουργέ, και να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την αντινάμωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόσμου. Του κόλπου, συγγνώμη. Είναι σημαντικό αυτό για τις μελλοντικέ μας σχέσεις και την γενικότερη συνεργασία στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αραβικά. Εάν θέλετε να φορέσετε τα ακουστικά σας. Στο όνομα του Ελέημονος και Μεγαλοπαπούς Θεού, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Εξωτερικών Αποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, η ειρήνη, το έλεος και η ευλογία του Θεού να σας συνοδεύουν. Θα ήθελα να εκφράσω την Μεγάλη τιμή που αισθανόμαστε για τι σχέσει συνεργασία, διαλόγου και διαβουλεύσεων που υπάρχουν μεταξύ του κράτου του Κατάρ και των διαφορών θεσμικών οργάνων και των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να εκφράσω ξανά το ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να ενδυναμώσουμε τέτοιου είδου σχέσει σε περιφερειακέ και διεθνεί διαστάσει. Επίση, ε, σκοπεύουμε να συνεργαζόμαστε στενά και να διαβουλευόμαστε για θέματα όπως αυτό της Λιβύης πρόσφατα, της Σομαλίας ή της Συρίας για να μην πω την τραγωδία της Συρίας, που αποτελούν παραδείγματα συνεργασίας, τα οποία χαρακτηρίζουν τις σχέσεις της Ευρώπης με το Κατάρ και της Ευρώπης με τον αραβικό κόσμο γενικότερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση, να απευθυνθώ στην συνεδρίασή σας, στην ομάδα, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σχέση με το τι κάνει το Κατάρ για τι σημαντικέ αλλαγέ και τι διαφορετικέ μετατροπέ που λαμβάνουν χώρα στον αραβικό κόσμο, γνωστέ ω αραβική άνοιξη, άνοιξη των αραβικών λαών. Λαών που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να κερδίζουν τη ζωή του τίμια και να καθορίζουν το δικό του μέλλον. Όταν αντιμετωπίζει κανεί λαϊκέ εξεγέρσει, οι ηγέτε δηλαδή, θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι παρά τι διαφορετικέ ε, συνθήκε, η φύση των προβλημάτων και το επίπεδο ανάπτυξη τη κάθε χώρα απαιτούν ενεργές διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, ε, διάλογο με τον λαό προκειμένου να ακούσουν τις ε, ανάγκες τους και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στα θεμέλια πολιτικών νομιμότητας και με στόχο την ευημερία. Με την αρχή των ε, κινήσεων διαμαρτυρίας θεωρήσαμε στο Κατάρ ότι αν δεν υπάρξουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν δεν θα υπάρξει και πρόοδος ότι η πολιτική της άρνησης δεν είναι μια λύση και ότι θα πρέπει να έχουμε μια ε, πραγματική στροφή προ μεταρρυθμίσει με ουσιώδη διάλογο και σπηρελτώντα ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτου και κοινωνία. Εάν έχουμε μάθει κάτι από την πρόσφατη την παλιότερη ιστορία μα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μάταιο να αντισταθούμε στι λαϊκέ αυτέ κινητοποιήσει. εμεις οπως και άλλοι, έχουμε πιστήσει την προσοχή εδώ και καιρό ότι επίκειται έκρηξη του ηφαιστείου. Για να θυμίσουμε αυτή μας την προειδοποίηση, πολλές εκθέσεις ε, του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ε, για την αραβική ανάπτυξη ε, από τις αρχές του 2002 εφιστούν την προσοχή στην ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών διαφορετικών διχασμών, για, την, για το χάσμα στην κοινωνία μεταξύ ηγετών και πολιτών, για τις, τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματο, για τι δημογραφικέ προκλήσει και βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι 50% των Αράβων είναι κάτω τη ηλικία των 24. Άρα αντιμετωπίζουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασία για του νέου, ιδίω για του ανέργου από πανεπιστημίων. Εδώ μιλάμε για μια πραγματική ορολογιακή βόμβα Πραγματική και καλυμμένη ε, ανεργία. Εδώ επίση υπήρχε και το διευθυντικό πρόβλημα των ε, τομέων τη παραγωγή σε περιφερειακό επίπεδο. Πραγματικά οι περιοχέ τη υπέθρου πλήσαν ένα βαρύ τίμημα κατά τη μετατροπή που ε, τέσσερι τελευταίε τελευταίες δεκαετίες ε, είχαν γνωρίσει οι χώρες αυτές όπου υπήρξαν οι εξεγέρσει και λόγω της απουσίας ενός κράτους ε, με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Πράγματι, το κράτος είχε εγκαταλείψει τελείως από το ρόλο και το μόνο που εξυπηρετούσε ήταν τα αστικά κέντρα με μια αντιπαραγωγική οικονομία που βασιζόταν σε έναν ε, ανεξέλεγκτο οικονομικό καπιταλισμό, ο οποίος όμως στις αναπτυσσόμενες αυτές κοινωνίες δεν τέριαζε γιατί δεν παρήχε και το απαραίτητο κοινωνικό δίκτυο προστασία. Ε, υπήρχε έτσι λοιπόν έλλειψη πολιτική συμμετοχή και βεβαίω οι κοινωνίε μα άρχισαν να γίνονται αποκλεισμένε ε, και να μην επιτρέπουν την ανάπτυξη ενεργών δυνάμεων και τάσεων της κοινωνίας των πολιτών που σκοπεύουν την ανανέωση. Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης δεν μπορούσε να μείνει εκτός των αραβικών κοινωνιών και να απαγορεύεται σε αυτές οι πρόσβαση στην γνώση, την διαδικτύωση και την ελεύθερη μετακίνηση. Έτσι λοιπόν οι αραβικές επαναστάσεις είχαν σχέση και με τις επαναστάσεις των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης όπως το Facebook και το Twitter και επίσης με τα αραβικά οπτικοακουστικά μέσα ή τα τηλεοπτικά κανάλια του αραβικού κόσμου τα οποία διδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων, στην παρακολούθησή του και βεβαίω έδειξαν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και δέσμευση ε, στην κοινότητα των αραβικών μέσων. Εδώ μιλάμε για τι επαναστάσει για την μεταρρύθμιση, γιατί εκπροσωπούνται ευρύτεροι τομεί, ε, περιφέρειε, τάσει και ηλικιακέ ομάδε, ακόμα και αν οι νέοι πάντοτε βρισκόνταν στο, στην πρώτη γραμμή. Οι νέοι πάντοτε ε, είχαν στόχο την αλλαγή την ίδια την αλλαγή που οι αρχές δεν είδαν να έρχεται ή δεν άκουσαν να χτυπάει την πόρτα μας, διότι κόφευαν και εθελοτυφλούσαν από πολιτικής σκοπιάς. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα ήθελα να τονίσω το βασικό γεγονός ότι παρά τις κοινέ πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές ε, σχέσεις των αραβικών λαών, τις ομοιότητές τους, τα κίνητρα και τα πρότυπα αλλαγής που πολλοί έχουν αποδεχτεί, Παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες σε κάθε κοινωνία. Πρώτα απ' όλα ε, εσωτερικοί παράγοντες οι οποίες ε, τον κανονίζουν το την δομή των κοινοτήτων, τη σύνθεσή του και τι συνιστότητε του. Και από την άλλη άποψη, ε, σημαντικό ρόλο παίζει η γεωστρατηγική θέση κάθε κράτου, ανάλογα με το πώ διαμορφώνεται και η εργατική του δύναμη, ο στρατηγικό του ρόλο. Κάτι που μπορεί να περιπλεκεί περισσότερο, ε, εφόσον οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί αυτοί παράγοντε μπορεί να συμπίπτουν. Η σημερινή κρίση στη Συρία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη δια σύνθεση τη κοινωνία. Κυρίε και κύριοι, από την αρχή των Αραβικών Επαναστάσεων, το Κατάρ έχει διδραματίσει ενεργό ρόλο στο να εξυπηρετεί και να διευκολύνει όσο το, δυνατότερο, όσο το δυνατόν περισσότερο την κατήρηση τη ειρήνη και προκειμένου να ε, περιορίσει τι αρνητικέ επιπτώσει. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στην ε, Ισία και αργότερα στην Αίγυπτο και εφόσον αυτά προχώρησαν λόγω των γετεροτήτων των δύο αυτών χωρών με, με πιο ταχύ ή πιο βραδύ ρυθμό, είδαμε ότι στην κρίση στην Ιεμένη τα πράγματα κινδύνευσαν να ξεπεράσουν τα εθνικά σύνορα. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου όρισε έναν οδικό χάρτη ώστε οι χώρες αυτές να ξεφύγουν από την κρίση αυτού του είδους. Το πρότυπο της επίλυσης κρίσης στην Ιεμένη είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα για να επιχειρήσουμε κατά ανάλογο και στη Συρία, λαμβάνοντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης υπόψη. Στην περίπτωση της Λιβύης, παρόλα αυτά, από την αρχή στο πλαίσιο του συνδέσμου των αραβικών κρατών, προσπαθήσαμε να προλάβουμε την επιδείνωση της κρίσης και να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ώστε ε, η ε, λιβική ηγεσία να υποχρεωθεί να δεχτεί την αλλαγή που ερχόταν έτσι να μην ε, οδηγηθεί η Λιβύη σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Η διπλωματία του Κατάρ μαζί με τις ε, αδελφές αραβικές χώρες και τις φίλες ευρωπαϊκές ε, χώρες Νομίζω ότι εδώ τήρησε μια θέση ιστορικής σημασίας Και τη λέω ιστορικής σημασία, διότι μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή στο ρόλο του αραβικού συνδέσμου και τι ευθύνε που αναλαμβάνει σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη. Εδώ ανέστηλε την συμμετοχή της ε, Λιβύης σε διάφορα όργανα του και βεβαίως αυτή περί λύση επαναλήφθηκε και στην περίπτωση της Συρίας όταν για εσωτερικούς λόγους ανεστάλλει η συμμετοχή αυτού του κράτους στον Αραβικό Σύνδεσμο. Έτσι Αναγνωρίστε στην περίπτωση τη Λιβύη ότι ο ρόλο του Αραβικού Συνδέσμου ήταν καθοριστικό, εφόσον εγκρίθηκε και το ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλεία το 1973, το οποίο ε, οδήγησε στη σωτηρία του λιβυκού λαού και έφερε τι απαραίτητε αλλαγέ. Κυρίε και κύριοι, σήμερα είμαστε μάρτυρε μια ανθρώπινη αραβική τραγωδία τεράστιων διαστάσεων, όπου το καθεστώ τη Συρία συνεχίζει να ε, χρησιμοποιεί στρατιωτικέ ε, λύσει και πολιτικέ προκειμένου να ε, ανακαιτήσει τις απαιτήσει για αλλαγέ από όλε τι συνιστώσει και τι μερίδε του Συριακού λαού. Θα ήθελ, έχω εδώ την τιμή να προεδρεύω στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Συρία που έχει δημιουργηθεί στο επίπεδο του Αραβικού Συνδέσμου. Μαζί με το Γενικό Γραμματέα και του Υπουργού είχα πάρα πολλέ επαφέ με την ηγεσία τη Συρία και του παρότρινα να σταματήσουν τι πράξει βία. Ο Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών έχει οθετήσει μια σειρά ψηφισμάτων και έχει διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη προκειμένου να, να επιληθεί αυτή η κρίση και έχει εκδιπλώσει ε, μια αποστολή, έχει δημιουργήσει μάλλον μια αποστολή παρατηρητών η οποία ξέρουμε τι τύχη είχε. Επαναλαμβάνουμε εδώ και πολύ καιρό και θα συνεχίσουμε να, να επαναλαμβάνουμε ότι η λύση θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια αραβικής πρωτοβουλία και ότι κάθε καθυστέρηση ή το να κλείσουμε και να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα θα φέρει περισσότερε επιπλοκέ. Η δολοφονία πολιτών δεν είναι λύση και βεβαίω κάποια από τα κόμματα δεν μπορούν να δώσουν λύσει στην κρίση του Συριακού καθεστώτο. Η Συριακή κυβέρνηση πιστεύει ότι και Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι υπάρχουν πράξεις τρομοκρατίας εναντίον της, πράξεις βίας ε, και γι' αυτό έχει ανατρέξει στις στρατιωτικές λύσεις. Όμως ε, το αντίθετο συμβαίνει, γιατί οι αριθμοί των θανάτων μεταξύ παιδιών που ξεπερνούν τι εκατοντάδε δεν μπορεί να σημαίνουν ότι τα παιδιά είναι τρομοκράτε, όπω επίση είναι πολλοί οι πολίτε οι οποίοι καταφεύγουν στην αυτοάμυνα για να μην χάσουν τη ζωή του, να μην φυλακιστούν ή να μην βασανιστούν. Η κυβέρνηση της Συρίας ε, λέει ότι κάποια κράτη-μέλη ε, αναπτύσσουν εναντίον της ε, μια, μια κρυφή ατζέντα. Αυτό όμως δείχνει ότι η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να έχει οθετήσει τέτοια στάση εφόσον όλοι έχουν καταδικάσει τέτοιε πράξει βία κράτη, ε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και οι ανθρωπιστικέ οργανώσει, οι οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν καταφύγαμε στο Συμβούλιο Ασφαλεία προκειμένου να βρεθεί μια λύση μέσω τη Αραβική Πρωτοβουλία, να αποσταλεί ένα διεθνέ μήνυμα και να στηρίξουμε την αραβική θέση προκειμένου να το καταλάβει αυτό το συριακό καθεστώ. Είπαμε ότι φτάνει ω εδώ, θα πρέπει να δούμε τι ζητά ε, ο Αραβικό και ο συριακό Λαό. Όμω, αντιμετωπίσαμε το βέτο τη Ρωσία και τη Κίνα. Ο, ο κόσμος ε, οθέτησε μια, έναν οδικό χάρτη και τα πλαίσια του σκοπό έχουν να βγάλουν τη Συρία από, αυτό το σκοτεινό, από τη σκοτεινή σύραγγα στην οποία έχει περάσει και στο επίπεδο τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη συνάντηση των φίλων του Συριακού λαού στην Τίνιδα, οι διεθνεί διπλωματικέ δυνάμει, σκοπό είχαν να περάσουν ένα μήνυμα προ τα κόμματα τη χώρα για να βοηθήσουν το καθεστώ, δηλαδή να ε, διατηρήσουν τη σταθερότητα και την ειρήνη εφόσον δυνατόν, αποφύγουν περισσότερου θανάτου μεταξύ των πολιτών και την αιματοχυσία και να διατηρηθεί το κράτο τη Συρία και η κοινωνία τη ε, στην εδαφική του ακαιρεότητα και την κυριαρχία του. Κάτι στο οποίο ανέκαθεν δεσμευόμασταν και αυτό εφόσον γίνει αποδεκτή η πρωτοβουλία του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και βασιζόμενη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου του Αραβικού Κόσμου 22 Ιανουαρίου 2012 και 12 Φεβρουαρίου 2012. Θα ήθελα εδώ να τονίσω την ανάγκη να αποσταλούν στα τεύματα κοινά των Αραβικών Κρατών και του ΟΗΕ προ τη Συρία, ώστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσουμε στήριξη στο λαό αυτό και να ε, υπάρξει η απαραίτητη ε, συνδρομή από ανθρωπιστικής πλευράς και για την αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών. Στόχος μας όλη αυτή την προσπάθεια είναι να σταματήσει η αιματοχυσία και να σώσουμε τη Συρία με τελικό στόχο, κάτι που έχουν εκφράσει όλε οι συνιστώσει τη Συριακή Αντιπολίτευσης, να ε, θεμελιωθεί μια δημοκρατία η οποία να κάνει σε τα δικαιώματα όλων. Η απόπειρα του καθεστώτο τη Συρία, να υποδαβλήσει φόβου ότι οι αλλαγές καθεστώτο της Συρία μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι κάτι το οποίο αντιφάσκει με την πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπο του ε, Εθνικού Συμβουλίου στο λόγο του στην Ισία ε, είπε ότι η αντιπολίτευση έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ότι η μεταχείριση των πολιτών της Συρίας είναι βάση του κατά πόσον έχουν την υπηκότητα ή όχι και τίποτε παραπάνω. Αυτό το αναγνώρισε ε, σαφώ το Εθνικό Συμβούλιο στη Συρία. Κυρίε και κύριοι, ε, οι προκλήσει τη Αραβική Άνοιξη είναι και εδώ δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο κόσμος μας αποτελεί ένα διεθνές χωριό. Το είδαμε στη Μεσόγειο θάλασσα, το είδαμε στον κόλπο ε, και καταλαβαίνουμε ότι το, ε, το συμβαίνει σε ένα σπίτι του χωριού επηρεάζει όλους ε, σε μια χρονική στιγμή. Είναι ένα πολύ, ε, υπάρχει ένα ακόμη πολύ σημαντικό ε, ζήτημα, το οποίο ήθελα να θίξω για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πολιτικού σκηνικού μπροστά μας. Νομίζω ότι τον εργαστούμε υπέρ της ε, μεταρρύθμισης μπορεί να μην οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, εάν δεν επιληθεί και το ζήτημα της Παλαιστίνης και αν δεν επιστρέψει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. Εάν αυτό το καθοριστικό ζήτημα δεν επιληθεί ή όλη η όλη γεωγραφική περιοχή θα παραμείνει σε κατάσταση ένταση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Ας περάσουμε αμέσω στη συζήτηση. Ο κύριος Αλαφράνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κασο κύριε Πρωθυπουργέ, εξ ονόματο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας, είναι πιστό σύμμαχος η χώρα σα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αραβική Άνοιξη και έπαιξε σημαντικό ρόλο και ε, εξακολουθεί να παίζει στην περιοχή, στο Λίβανο, στην Ερυθρέα και αλλού. Είστε και βασικός ε, συνεισφορέας στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία και ε, το ε, πρόσφατο ψήφισμα δεν ήταν δεσμευτικό για τη Συρία σε ένα όργανο που εσείς προεδρεύετε. Ποια είναι η κατάσταση στο Ιράν και η σχέση σας με τη Συρία. Να ρωτήσω πρώτα για τη Συρία. Εσείς θέλετε να εκδοθεί ένταλμα για το Διεθνές Δικαστήριο ε, εις του Πρόεδρου Άσατη. Όπως είπε ο υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια. Καταλαβαίνετε τι εννοεί. Στην υποστήριξη της ε, αντιπολίτευσης και των αντιφρονούντων στη Συρία. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αναλύετε την κατάσταση στο Ιράν και πώς αντιμετωπίζετε το θέμα των πυρηνικών όπλων εκεί και πώς σας φαίνονται τα τύμπονα του πολέμου που ακούγονται στον ορίζοντα στην περιοχή. 17 διμερείς συμφωνίες έχετε με 17 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αεριακή κυκλοφορία και ξέρω ότι είστε σε διαπραγματεύσεις με άλλες πέντε χώρες και είστε σε επαφή με τον ε, Επίτροπο Αρμόδιο για την ε, αέρια κυκλοφορία και θέλετε να κάνετε μια συμφωνία ε, ελευθέρων ουρανών ανοιχτών εθέρων. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κυρία Γκόμες. Χαίρετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λιβύη, εκτιμώ πολύ το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα σας στην απελευθέρωση της Λιβύης από τη δικτατορία, τη στιγμή δικτατορία που ζούσε, ίσως στιγνότερη από άλλες. Εκτιμώ επίσης και το ρόλο της χώρας σας ε, που φιλοξενεί το κανάλι Al Jazeera, που είναι σημαντική πηγή πληροφορίας και ενημέρωσης όχι μόνο για τον αραβικό κόσμο, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Μ' αρέσει πολύ η Al Jazeera. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχω εδώ μια έκθεση της Freedom House που αναφέρεται στα περσινά γεγονότα καθ' όλη τη διάκρια του έτους και αναλύει τις πολιτικές ελευθερίες και τις δημόσιες ελευθερίες και ταξινομεί τις χώρες. Τη χώρα σας την κατατάσσει ως ανελεύθερη χώρα. Λίγο πιο πάνω από το Ιράν. Δύο θέσεις πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί όλες αυτές οι σημαντικές ιδέες που μόλις μας παρουσιάσετε για τον τρόπο που καταλάβατε πώς ε, ε, κρύγνεται αυτό το ηφαίστειο. Όλα αυτά δεν μπορούν να μεταφραστούν στη χώρα σας και στο λαό σας και εκείνους που φιλοξενείτε όπως είναι οι μετανάστες εργαζόμενοι και οι γυναίκες φυσικά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, σε σχέση με τη Λιβύη σημείωσα συγγνώμη, το πολύ σημαντικό ρόλο σας αλλά άκουσα ότι υπάρχουν και κάποιες τάσεις ακραίων φαινομένων που υποστηρίζονται από ε, πολίτες του Κατάρ. Υποστηρίζουν ακραία στοιχεία που στο μέλλον ε, μπορεί να οδηγήσουν και σε νέα έκρηξη φυστίου. Για τη Συρία λοιπόν, επίσης, πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε να ενωθεί η αντιπολίτευση που φαίνεται τόσο κατακαιρματισμένη γιατί μιλήσατε για ε, τραγωδία και ε, για το μέλλον. Πώς μπορεί να βοηθηθεί εκεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Uh, ε, Mr. President. Η κυρία Νέιτς, ε, Πρόεδρε, συνάδελφε, κύριε Πρωθυπουργέ, εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Είχα τη χαρά να είμαι προσκεκλημένη στη χώρα σας ε, πριν από 10 χρόνια και πλέον κατά τη διάρκεια της υπουργική διάσκεψης που οδήγησε στη Συμφωνία της Δόχα για το Παγκόσμιο Εμπόριο και τον ΠΟΕ. Ήμουν λοιπόν ε, σε θέση να απολαύσω τη φιλοξενία σας και με χαρά σας καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο. Όπως ε, ανέφερε και ο συνάδελφος Αλαφράγκα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το Ιράν όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις παλιές μας ανησυχίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και όλες τις εκθέσεις για την αυξανόμενη καταστολή του πληθυσμού, ιδιαίτερα εν ώψη των επικείμενων εκλογών και όσων θα επακολουθήσουν. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη. Ποια είναι η άποψή σας για την εξελίξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Γι' αυτό επηρεάζει γενικά τα ενεργειακά τιμολόγια στην παγκόσμια οικονομία. Σας ευχαριστώ. κυρία Φλότρο. Ζητώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι μου είχατε δώσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Εγώ θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε τη στρατηγική σας και τη σκέψη σας στη Συρία. Εδώ είμαι, στα αριστερά σας. Σας βλέπω, απλώς ζήτησα τα γυαλιά μου να μου φέρουν. Α, για να με βλέπετε καλύτερα. Μάλιστα, περιμένω. <laughs> Euh, je voulais vous inviter donc θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω κύριε Υπουργέ να διευκρινίσετε πιο συγκεκριμένα ε, ποια είναι η στρατηγική σας σε σχέση με τη Συρία. Γιατί γνωρίζετε ότι οι φίλοι της Συρίας την είδα δεν κατέληξαν σε ένα ψήφισμα που να περιλαμβάνει τα όσα εσείς είπατε. Δηλαδή ανάπτυξη ε, δύναμη του ΟΗΕ ε, με ε, συμμετοχή Αράβων στη Συρία. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και οι προπτικές και για τους ε, λεγόμενους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Δηλαδή κάποια στιγμή, εκτός αν αποφασίσει κάποιος να συγκρουστεί άμεσα με τον Άσαντ, να επιτύχουμε να σταματήσει ε, τις εχθροπραξίες. Δεν ξέρω πώς θα το επιτύχουμε και αν συμφωνείτε. Ε, μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Ρωσία, να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Ε, αυτός ο δρόμος είναι αξιόπιστος, είναι σοβαρός. Αυτό έχει υπόψη σας. Αλλιώς πώς φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν οι δυνάμεις εκεί να αναπτυχθούν στη Συρία στρατεύματα χωρίς να είμαστε σε εμπόλεμη σύραξη ή ένα σενάριο τύπου Λιβύης. Θα σας παρακαλούσα λίγο να το διευκρινίσετε διότι θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πραγματικά αφόρητη πλέον και δεν βλέπουμε τις στρατηγικές επιλογές ε, που θα είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι από εκείνους που είχαμε αντισταθεί με κάθε τρόπο στην ε, νατοϊκή επέμβαση και στον πόλεμο στη Λιβύη και νομίζω ότι έχουμε δικαιωθεί από τις εξελίξεις δεν πιστεύω ότι ο κύριος Πρωθυπουργό πιστεύει τα όσα λέει για τα προβλήματα της νεολαίας και των κοινωνιών στον αραβικό κόσμο και στη χώρα του. Διότι αν πίστευε αυτά τα πράγματα δεν θα ε, είχε η χώρα την οποία αντιπροσωπεύει και η κυβέρνηση μια τέτοια επιθετική, ιμπεριαλιστική πολιτική που βοηθάει τον ΝΑΤΟ και τις δυνάμεις σε έναν ανταγωνισμό για, τα, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτά που υπόθηκαν για τα κοινωνικά προβλήματα τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη, αλλά δεν φαντάζουμε ο κύριος Πρωθυπουργό να στέλνει τις δυνάμεις του Κατάρ και στην Ελλάδα, ας πούμε, για να τακτοποιήσει την κατάσταση. Να είμαι τώρα πιο συγκεκριμένο, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπάρχουν δημοσιεύματα του BBC που λένε ότι η χώρα σας είχε ήδη πριν την ε, ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του πόλεμου του ΝΑΤΟ στην ε, Λιβύη 7.000 στρατιωτικούς στη Βενγάζη. Αυτή η πληροφορία δεν διαψεύτηκε ποτέ, τουλάχιστον δεν την έχω υπόψη μου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εγώ και άλλοι πιστεύουμε ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι πραγματικά η για τη δημοκρατία για την απελευθέρωση των ε, λαών από δικτάτορες, που όντως ο Καντάφη ήταν τέτοιος δικτάτορας, ή μήπω υπάρχουν άλλου είδου βλέψει που η χώρα σα έχει γενικότερα στην περιοχή. Δεύτερον, με τα ζητήματα αυτά, με τα δεδομένα αυτά θέλω την ε, άποψή σα για το πόσου στρατιώτε αυτή τη στιγμή το Κατάρ έχει στη Συρία και πότε ετοιμαζόσαστε να επέμβετε ε, στο ε, Ιράν. Μου κάνει επίση τεράστια εντύπωση η, η θεώρηση των πραγμάτων που έχετε για τι εξελίξει στη Συρία που τουλάχιστον για λόγους ισορροπία θα έπρεπε κανεί να, περιμένει και τη γνώμη της άλλης άποψης και της άλλης χώρας. Δεν είσαστε μόνο εσείς στη Συρία και δεν είσαστε μόνο εσείς που δρείτε εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε, είμαι πάρα πολύ ανήσυχο, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι σας άκουσα να μιλάτε για στρατιωτική επέμβαση του συνδέσμου των αραβικών κρατών στη Συρία, αφήνοντας κατά μέρο πια και επίσημα τα όσα κατά καιρού η χώρα σας έλεγε για το διεθνές δίκαιο, για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, εάν η χώρα σα συνεχίσει αυτή την πολιτική και μου κάνει εντύπωση, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί από όλε τι χώρε του Συμβουλίου Συνεργεια του Κόλπου, ειδικά το Κατάρ, έχει μια τέτοια επιθετική πολιτική. Μια τέτοια επιθετική πολιτική η οποία βέβαια δεν έκανε τίποτα για το θέμα των Παλαιστινίων στη Γάζα. Μα είπατε κάτι στο τέλο, αλλά αυτά είναι λόγια του αέρα. Δεν σα είδαμε να είστε τόσο αποφασισμένοι για το θέμα του Παλαιστινιακού λαού. Λέω πάλι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η χώρα σας είναι τόσο επιθετική στα πλαίσια του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και παραδείγματος χάρη εσείς οι ίδιοι συμβάλλατε στην καταστολή της λαϊκής εξέγερσης στο Μπαχρέιν. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση. Τέλος, θέλω μια άποψη ε, τι θα κάνετε εάν τελικά ο εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, κατηγορήσει δυνάμεις του, του Κατάρ για εγκλήματα πολέμου στη Λιβύη, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μου βέβαια, ε, για εγκλήματα πολέμου του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στάνοκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω θερμά τον Πρωθυπουργό ε, Φενή από την ομάδα μου ε, των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Μόλις έρχομαι από μια συνέντευξη ε, και σας συγχαίρω για την Al Έχει γίνει παγκόσμιο κανάλι ε, ε, εδρεύει στη Δόχα και την υποστηρίζει και ε, η κυβέρνησή σας. Το Κατάρ είναι πρωταγωνιστή στον αραβικό κόσμο και στο Συμβούλιο Συνεργασίας του ε, Περσικού Κόλπου. Εγώ προβληματίζομαι λίγο για το ρόλο που θέλετε να παίξετε στις εξωτερικές σχέσεις. Είστε πλούσια χώρα πλην μικρή, με λίγο πληθυσμό και λίγες ένοπλες δυνάμεις, περιορισμένες και βλέπουμε στην ε, Αρινή Άνοιξη, στην ε, Αραβική Άνοιξη, συγγνώμη, ε, τους λεονταρισμούς σας λίγο. Μέχρι και όπλα στείλατε στη Λιβύη και τελικά έπεσαν στα χέρια των Ισλαμιστών. Και τώρα τα πουλάνε στην Αλκάιτα, στο Σαχέλ. Και είναι λυπηρό αυτό, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η στρατηγική σας θεώρηση και το όραμά σας για την περιοχή. Θέλετε περισσότερη δημοκρατία, υπάρχει ανάγκη εκεί. Εγώ ανέκαθεν πίστευα ε, στις ε, γνήσιες μοναρχίες της Μέσης Ανατολής σε σχέση με τις ψευδομοναρχίες τύπου Κοεντάφη, Μουμπάρακ και Οικογενοκρατίες. Οι δικές σας μοναρχίες, ε, μοιράτα του κόλπου, συνταγματική μοναρχία ε, είναι το μέλλον σας ε, σαν την Ιορδανία ή το Μαρόκο. Πώς φαντάζεστε τη μετεξέλιξη της περιοχής σας συγκεκριμένα και γενικότερα της Αραβικής Άνοιξης. Γιατί πολύ γρήγορα γίνατε πρωταγωνιστής, ενώ ξεκινήσατε πολύ ταπεινά και σεμνά και χαμηλά και ξαφνικά αναρωτιέμαι γιατί αυτή η κυριαρχία στη διεθνή σκηνή. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αραβικά. και να κατηγοριοποιήσω τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. κατά Αρσυρία, Λιβύη, ε, με θεματικές ενότητες έτσι για να καλύψουμε όλα τα θέματα και τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στη Συρία και στην κατάσταση εκεί. Αυτή τη στιγμή εμείς ως διεθνής κοινότητα ε, κρατών θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας και στις υποχρεώσεις μας. Θα πρέπει να προεξοφλήσω ότι το Κατάρ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αναμειχθεί στην εσωτερική κατάσταση οποιασδήποτε άλλης χώρας και στις εσωτερικές υποθέσεις. Ούτε συμφέροντα έχει ιδιαίτερα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Γνωρίζετε ότι το Κατάρι είναι ένα κράτος πλούσιο, πλην ε, μικρό. Έχει όμως και φιλοδοξίες για τη σταθερότητα της περιοχής. Δηλαδή, θέλουμε να επιληθούν ειρηνικά όσο γίνεται οι θερμές αιστείες στην περιοχή μας. Είτε είναι το Ιράν, είτε είναι η Συρία, είτε το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Ακόμα και η Βόρειος Αφρική. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κρίσεις που χρειάζονται διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπιστούν και άλλες κρίσεις που χρειάζονται περιφερειακή συνεργασία. Ε, τα αραβικά κράτη, ας πούμε, ε, μαζί με τη διεθνή κοινότητα. Για τη Συρία και για τη Λιβύη. Πρέπει να πω ότι το Κατάρ γεωγραφικά απέχει πάρα πολύ από τη Λιβύη. Ε, αλλά όταν είδαμε ότι υπάρχει ένα κράτος όπου ο αρχηγός κράτους άρχισε να στέλνει αεροπλάνα, πυράβλους, τάγκς απέναντι στον ανυπεράσπιστο λαό του και μέσα σε δύο ώρες έχασαν τη ζωή του στη φυλακή Αμπουσλίν πάνω από 1.200 κρατούμενοι. Όταν είδαμε ε, τις ε, όταν είδαμε το καθεστώς τη μεταχείριση επιφύλαση στο λαό του, σε ένα λαό που είχε εξεγερθεί ειρηνικά, αναμίχθηκε όντως το Κατάρ για να προστατεύσει το λιβικό λαό. Είπε κάποιος ότι είχαμε 7.000 στρατιωτικούς προηγουμένως ήδη στη Βενγάζη. Αλλά ο πληθυσμός του Κατάρ και τα στρατεύματά μας δεν φτάνει. Εμείς δεν έχουμε 7.000 ε, στρατό να μπορέσουμε να στείλουμε εκ των προτέρων στη Βενγάζη. Εκ των υστέρων, μετά τα γεγονότα, στείλαμε μερικά στρατεύματα εκεί για ανθρωπιστική βοήθεια και όταν αποφασίστηκε ε, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ να ε, γίνει μια συμμαχία για να σώσουμε το λιβικό λαό και να αποτρέψουμε να σταματήσουμε την αιματοχυσία στη Λιβύη. Γιατί η αιματοχυσία ήταν πριν επέμβει το ΝΑΤΟ. Όταν ελήφθη η απόφαση αυτή στο Παρίσι, είχαμε δύο τεινά μπροστά μας ως διεθνής κοινότητα κρατών στην οποία διεθνή κοινότητα ανήκουμε κι εμείς. Ή θα αφήναμε τη Βενγάζη τελείως απ' έξω ε, ή θα επεμβαίναμε. Ο Σαΐφ Αλ Ισλάμ είχε πει στο Συμβούλιο Ασφαλείας μάλλον πριν πάρει η απόφαση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα είχαν ισοπεδώσει τη Βενγάζη. Το είχε δηλώσει αυτό ο Σαΐφ Και τότε αποφασίσαμε να επέμβουμε. Και άρχισαν οι ε, δράσεις διάσωσης για να σώσουμε πραγματικά το λιβικό λαό. Και ήταν ε, μεγάλη η διεθνής συμμαχία. Τι συμφέροντα έχουμε. Δεν έχουμε συμφέροντα στη Λιβύη ούτε πριν ούτε μετά. Το Κατάρ έχει περισσότερο πλούτο από τη Λιβύη. Έχουμε αρκετό πλούτο στη διάθεσή μας. Και το Κατάρ έχει πληρώσει και πανάκριβα τη διάσωση αυτή του λιβικού λαού. Μετά από 40 χρόνια καταστολής και καταπίεσης. Εμείς σεβόμαστε όλους τους Λιβύους, αλλά πραγματικά το καθεστώς ήταν γελίο. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη μεταχείριση αξίζει σε ένα τέτοιο καθεστώς. Υπήρξαν και διεθνείς συνέπειες από το καθεστώς αυτό. Θυμάστε τις αεροπηρετίες, τα, ε, τις εκρήξεις βομβών και ε, τις καταρρύψεις αεροσκαφών. Έπρεπε να τερματιστεί αυτό το καθεστώς. Ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει αυτή τη δικτατορία όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό και δια της βίας μάλιστα σε άλλες χώρες. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Λιβύη δεν είναι ικανοποιητικά. Φυσικά, ορισμένοι αναφέρθηκαν σε Ισλαμιστικές ομάδες. Κοιτάξτε, εσείς είστε δημοκρατικοί λαοί. Ε, εκπροσωπείται όλους τους λαούς της Ευρώπης και εμείς ε, σεβόμαστε την επιλογή των Ευρωπαίων και των πολιτών να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους. Στην Τινησία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο δεν θα πρέπει να εκλέγονται οι εκπρόσωποι από τους λαούς, δεν θα πρέπει να τους σεβόμαστε. Αυτό που χαρακτηρίστηκε η Ισλαμιστική κυβέρνηση και οι φόβοι που υποδαβλίζονται δεν είναι σωστό. Αυτοί προέρχονται από την κοινωνία. Ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Δεν το γνωρίσαμε ποτέ αυτό το καθεστώς. Ας δούμε. Σέβονται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ανταποκρίνονται στο καθήκον τους, εκπροσωπούν τους λαού του. Εάν το επιθυμούν αυτό οι λαοί, εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε τις επιθυμίες των αραβικών λαών. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων και οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε και να τη σεβόμαστε. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε μια κυβέρνηση αν είναι Ισλαμιστική ή όχι. Θα πρέπει να σεβόμαστε κάθε κυβέρνηση που εκπροσωπεί το λαό τη και ανταποκρίνεται και σέβεται στι επιθυμίες του λαού. Για τον υπερελισμό και το τι συμβαίνει στη Συρία τώρα. Εμείς ανέκαθεν είχαμε καλές σχέσεις με τη Συρία, αλλά αν πρέπει να επιλέξουμε το λαό ή την εξουσία, θα επιλέξουμε το λαό της Συρίας. Γιατί ο λαός είναι αυτός που θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Δεν μας ικανοποιούν τα όσα συμβαίνουν στη ε, Συρία. Δολοφονίες, ε, ε, θάνατοι γυναικών, παιδιών. Εμείς θελήσαμε να παρέμβουμε στη Συρία με ειρηνικό τρόπο. Προσπαθούμε έξι μήνες ολόκληρους και παραπάνω από έξι. Εδώ και ένα χρόνο γενικότερα ε, προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα αυτά εντός του αραβικού οίκου, αλλά δεν τα καταφέραμε, διότι το καθεστώς στη Συρία δεν θέλησε να δεχτεί την αραβική λύση. Στείλαμε παρατηρητές στη Συρία. Για πρώτη φορά ο Αραβικός Σύνδεσμος πράττει κάτι τέτοιο, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε λύση. Διαπιστώσαμε ότι γίνονται προσπάθειες να αποκρυ ακολουθούν διάφορα τεκτενόμενα ε, να κολλησιεργήσουν, προσπαθούν ε, να λύσουν τα πράγματα μόνοι τους. Ο Συριακός λαός αξίζει περισσότερα από μας και όχι αυτές τις ε, χρονοτριβές και τις κολλησιεργίες. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη σύγκρουση. Πολύ ωραίο θα ήταν να μπορέσει κανείς να βρει ειρηνική λύση που να δέχεται και ο λαός της Συρίας, κυρώσεις ας πούμε. Έχουν δείξει όλες οι εκθέσεις όμως και ε, τα γεγονότα ότι δεν μπορούμε να βρούμε ειρηνική λύση. Έχουν αρχίσει βομβαρδισμούς τώρα από αεροπλάνα. Είδαμε ότι επί δέκα μήνες η επανάσταση αυτή ήταν ειρηνική. Παρόλα αυτά, παρόλες τις διεθνείς προσπάθειες, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε τις εξελίξεις. Η αυτοάμυνα είναι και νόμιμη και θεμητή. Όταν άρχισε ο λαός με πολύ περιορισμένα μέσα να προσπαθεί να προστατευτεί, τους χαρακτήρισαν τρομοκράτες. Τα γνωστά πάντα προσπαθεί κάποιος ε, να ε, τους ε, προσάψει ότι είναι μέλη της αλκαϊδα Και εδώ στην Ευρώπη, μόλις ακούσουν Αλκάιντα, αρχίζουν να ενδιαφέρονται. Υπάρχουν στη Συρία Ισλαμιστές και μουσουλμάνοι. Εγώ είμαι περήφανο που είμαι μουσουλμάνος, αλλά μουσουλμάνος δεν σημαίνει τρομοκράτη αυτόματα. Οι μουσουλμάνοι ε, στη Συρία είναι ίδιοι με τους μουσουλμάνους στην Τουρκία. Δεν θα πρέπει να είμαστε εχθρικά διακείμενοι απέναντί τους. Στην Παλαιστίνη, Φερρυπίν, στη Γάζα, ε, εξελέγει ελεύθερα και δημοκρατικά μια κυβέρνηση από το λαό. Από τον Παλαιστινιακό λαό. Και παρόλα αυτά, την κυβέρνηση αυτή η οποία έχει εκλεγεί δημοκρατικά και ελεύθερα. Εσείς οι ίδιοι που είστε δημοκρατικά και ελεύθερα εκλεγμένοι δεν θελήσατε να τη δεχτείτε. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε στη Συρία θέλουμε επέμβαση. Και δεν ισχύει ότι ε, θέλουμε να στείλουμε στρατεύματα, ούτε έχουμε αυτή τη στιγμή στη Συρία. Δεν έχουμε σκοπό να καταστρέψουμε τη Συρία εμείς επιθυμούμε να δούμε πώς θα μπορέσει να ζήσει ελεύθερα ο Συριακός λαός, να εκλέγει ελεύθερα ε, τους εκπροσώπους, τους βουλευτές, την κυβέρνησή του, να ορίζει τις τύχες του. Είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων στη Συρία και οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν θα έρθουν με αερολογίες της κυβέρνησης και φρούδες, ελπίδες και υποσχέσεις. Εμείς θέλουμε ένα ειρηνικό πρόγραμμα. Δεν μιλάμε για στρατιωτική επέμβαση. Ειρηνική επίλυση για να επιτύχουμε αυτό που επιθυμεί ο Συριακός λαός. Το καθεστώς όμως αρνείται να ε, μπει σε αυτή την ατραπό. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την τρομακτική ανθρωπιστική κατάσταση πλέον στη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε διαφορετικό από το να στείλουμε βοήθεια. Δεν είναι σωστό να απαιτήσουμε να σταματήσουν αυτές οι καταστάσεις. Εμείς και ο Εμμύρης του Κατάρ ζήτησε και απέτησε να αποσταλεί ειρηνευτική δύναμη, αραβική και διεθνής, έτσι ώστε να ε, τερματιστεί η αιματοχυσία και να προωθηθεί μια ειρηνική επίλυση της κρίσης. Με πολιτικά μέσα. Αλλά η κρίση αυτή είναι τόσο βαθιά, απλούστατα, που δεν μπορούμε να τη λύσουμε συναισθηματικά με συναισθήματα και πάθη. Και... Λέτε να μην επέμβουμε στρατιωτικά. Ποιος το επιθυμεί και ποιος δεν το επιθυμεί. Ποια είναι τα συμφέροντα. Εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Συριακού λαού. Τα, τα συμφέροντα των υπολείπων έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά τα συμφέροντα του Συριακού λαού. Και ο Συριακός λαός αυτή τη στιγμή υποφέρει τα πάνδυνα. Πριν έρθω στο Ιράν όμως, θα ήθελα να πω ότι θα επιθυμούσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει περισσότερη και βαθύτερη κατανόηση για αυτά τα θέματα. Μην τα βλέπετε παρακαλώ μερός. Μην τα βλέπετε μόνο από το πρίσμα ενός κόμματος ή ε, μιας πλευράς. Είναι ανθρωπιστικό το ζήτημα. Θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε ε, πραγματικά ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Δεν θέλουμε να στείλουμε στρατεύματα στη Συρία να επέμβουν δια της βίας. Ε, ειρηνευτικά ε, στρατεύματα για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ζωές γυναικών και παιδιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει καθημερινά ε, την αιματοχυσία μπορείτε να το αφήσετε αυτό να διονύζετε. Απευθύνομαι στη συνείδησή σας. Δεν μπορεί να το δέχεστε αυτό. Δεν χρειάζεται καν συζήτηση τέτοιο θέμα. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε διάβγεια ε, στην ε, θεώρησή μας και όχι ομάδες συμφερόντων. Ξέρω ότι υπάρχουν λόμπι που έχουν διάφορα συμφέροντα και προσπαθούν να επηρεάζουν για να πείσουν και αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας συνιστώ να τα κοιτάτε όλα αυτά αντικειμενικά. Άλλα θέματα το Ιράν. Είμαστε κατά ιασδήποτε στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν. Επιθυμούμε ειρηνική λύση του θέματος. Το Ιράν είναι γείτονα του Κατάρ και σημαντικός εταίρος στην περιοχή. Εμείς επιθυμούμε διπλωματική λύση αυτού του ζητήματος. Θέλουμε να καταβληθούν προσπάθειες για τις διπλωματικές οδού για να βρεθεί μια λύση σε συνεργασία με το Ιράν. Διάλογος χρειάζεται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το Ιράν είναι μεγάλη χώρα και αποφασιστικός παράγοντας στην περιοχή μας. οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα πυρηνικό εργοστάσιο για ειρηνικούς σκοπούς και πολιτικούς σκοπούς. Εάν ισχύει αυτό, έχουν το δικαίωμα. Αλλιώς ας το εξετάσουμε. Εμείς είμαστε κατά της ε, πυρηνικής ενέργειας για μη ε, ειρηνική χρήση. Γιατί οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα οδηγούσε σε κούρσα πυρηνικών όπλων και εξοπλισμών στην περιοχή και αυτό είναι επικίνδυνο. Αλλά Είμαστε πεπισμένοι ότι η λύση θα πρέπει να είναι ε, μια λύση στην οποία να συμμετέχουν όλες οι χώρες της περιοχής για να ε, μπορέσει να λήξει αυτό το θέμα. Ορισμένα αναφερθήκατε στη χώρα μου. Το κατάρα. αυτό θα το αφήσω, τελευταίο ήθελα να το αφήσω. Πρώτον, δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι σωστά αυτά που αναφέρατε στην έκθεση για το κατά. Για τις γυναίκες ας πούμε, έχουμε γυναίκα υπουργό, έχουμε γυναίκες πρέσβης. Οι γυναίκες δραστηριοποιούνται σε, όλη, σε όλο το φάσμα της κοινωνίας στο κατά και σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ευθεριών και των δικαιωμάτων. Δεν έχουμε πολιτικούς κρατουμένους ας πούμε. Έχουμε σύνταγμα. Σύγχρονο. Και όλοι οι απολύτες ε, του Κατάρ αποφάνθηκαν σε δημοψήφισμα. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένα σύνταγμα που τους επέβαλε η κυβέρνηση ή ο Εμμύρης. Ήταν ένα σύνταγμα που θέλησε έτσι ο λαός. Ε, και δέκα χρόνια έχει τεθεί σε ισχύ και επίσης έχουμε και περιφερειακές εκλογές, ερετούς ε, εκπροσώπους, ε, δήμους, κοινότητες, περιφέρειες, ε, εμπορικό επιμελητήριο. Ε, πάλι ερετό, αναφερθήκατε στο τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera. Γνωρίζουμε ότι πολλοί στον αραβικό κόσμο και αλλού μας επιτίθενται λόγω του Al και λόγω του τύπου και της ελευθεροτυπίας στο Κατάρ. Και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται απολύτως σεβαστά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η έκθεση αυτή έχει εσφαλμένες προφορίες, γιατί ε, ο ΙΕ και άλλα διεθνή φόρα έχουν ε, κάνει εκθέσεις που λέγουν ότι έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στο Κατάρ. Του χρόνου, γι' αυτού η ψηλότης ο ε, Εμμύρης εξήγηλε ελεύθερες βουλευτικές εκλογές. Ε, θέλουμε πραγματικά το Κατάρ να εξελίσσεται κοινωνικά, οικονομικά, σε ε, σύμπνια πάντα με το Σύνταγμα για το οποίο ψηφίσαμε όλοι. Αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε και τις παραδόσεις μας, τις ε, Ισλαμικές παραδόσεις, τις Αραβικές παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα. Είναι καλοδεχούμενη κάθε επικοδομητική ε, κριτική ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια που στόχο έχουν να μας βοηθούν πάντα για να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Και ελπίζω... Αν, αν ξέχασα τίποτα ή αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλες τέσσερις ερωτήσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα λεπτό παρακαλώ έκαστος να περιοριστείτε για να προλάβουμε να απαντήσουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Ρωμέρο. Ευχαριστώ πρώτο. Ναι, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, Πρωθυπουργέ. Αξιολογούμε θετικά και εκτιμούμε τις προσπάθειές σας στον Αραβικό Σύνδεσμο για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Θέλω να σας ρωτήσω τι κάνετε για την υποστήριξη ε, στα σαλαφιστικά κινήματα. Έχετε ταμείο που διαχειρίζεται ποσά, είναι διαφανές και για ποια ποσά συζητούμε, τι τάξη μεγέθους. Δεν ναι, με βλέπετε εδώ, απέναντί σα είμαι. Ε, περί ποιων ποσών πρόκειται και πώς ελέγχετε εσείς αυτό το ταμείο. Γιατί οι σαλαφιστές είναι Ισλαμιστές, αλλά ε, συνδέονται με την τρομοκρατία και δεν ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζεται ε, σε σχέση με τις ένοπλες πολιτοφυλακές στη Λιβύη και την τη ρόλο παίζουν και στο Σαχέλ, στις ένοπλες ομάδες και πολιτοφυλακές. Θέλω συγκεκριμένα να σας αναφέρω ε, ε, το Πανεπιστήμιο της Αζεϊτούνα που κάνουν δικαστήρια, λαϊκά δικαστήρια, οι ίδιοι οι καθηγητές εκεί και αποφαίνονται πώς θα φερόμαστε στις γυναίκες, στα παιδιά μας, στην οικογένεια, τι θα κάνουμε. Ε, αυτοί ε, οι σαλαφιστές ε, χρηματοδούν από εσά και με ποιο τρόπο. Ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, θα κάνω συγχαρητήρια τα οποία θα απίφθηνα διαφορετικά στον Πρωθυπουργό για ε, τα επιτεύγματά τους διότι η Ντόχα έγινε ε, πολύ γρήγορα ένα κέντρο της παγκοσμίου πολιτικής και σας συγχαίρω και για την Αλτζεζίρα και για ό,τι αντιπροσωπεύει ένα παράθυρο προς την Ιφίλιο. Αλλά θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο. Πώς διαβλέπετε τις εξελίξεις της διαμάχης μεταξύ Ισραήλ και ε, Παλαιστίνης, διότι η λύση των δύο κρατών δεν φαίνεται φαίνεται όλο και περισσότερο σαν ε, να είναι ένα ευχολόγιο, μια φάτα μοργάνα των Ισραηλινών. Οπότε ε, τι μέλη με τις εκλογές της Παλαιστίνης. Θα πρέπει να τις σεβαστούμε. Θα ήθελα να τις σχολιάσετε. Και ε, ε, είχαμε την ε, παρέμβαση του JCC στο Μπαχρέιν σχετικά με τις, τα στρατεύματα της Σαουδικής Αραβίας στο Μπαχρέιν, πράγμα που δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης πίσω μιας τέτοιας κατάστασης. Κύριε ε, Πρωθυπουργέ, αναλύσατε τις αιτίες της Επανάστασης, Πώς όμως εσείς διαβλέπετε την ε, έκβαση διότι η ε, επαναστασή είναι μία ατελής διαδικασία αλλά αν πάρουμε την Αίγυπτο οι νέοι ε, θα ήθελαν περισσότερη ελευθερία και τώρα υπάρχουν περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι από ό,τι επί Μουμπαράκ και ήθελαν μία πιο εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και και τώρα η οικονομία καταραίει. Η ε, Αιγυπτός θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, οπότε πώς εσείς διαβλέπετε την κατάσταση ή στην Αίγυπτο και στον Μπαχρέιν όπως σας είπα διότι η επανάσταση διακόπηκε δια μίας επεμβάσεως Πώς λοιπόν αξιολογείτε την κατάσταση στο Μπαχρέιν και σας συγχαίρω βεβαίως όχι μόνο για τα επιτεύγματά σας στη Μέση Ανατολή, στα πλαίσια της διεθνούς διπλωματίας ε, και ε, στην διπλωματία αυτού του τόσο ε, προσφυλούς ενδιαφέροντος που έχουμε όλοι, δηλαδή του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, έχω και εγώ μία σύντομη παρέμβαση. Θα ακούσουμε Όλε όλες τις θέσεις και μετά θα διαμορφώσουμε την άποψή μας αλλά είμαστε πολύ ευγνώμοστες ότι εσείς και η χώρα που είναι τόσο σημαντική μας ε, μεταδίδετε αυτές τις πληροφορίες. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που ελέγχθη περί της ε, Αιγύπτου διότι εγώ στην ε, Αίγυπτο έχω την εντύπωση ότι η νεολαία του Twitter είναι η χαμένη στην αλλαγή αυτή και θα πρέπει και ότι γίνεται κάτι το οποίο μπορεί να μην δημιουργεί προβλήματα, αλλά ε, ε, τα υπόλοιπα ιδρύματα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και ε, ότι υπάρχουν παρεμβάσεις άλλων κρατών που χρηματοδότησαν τις εκλογές στην Αίγυπτο και δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια πλουραλιστική εξέλιξη. Δεύτερη ερώτηση βάσει τη εμπειρίας στην Αίγυπτο. Στη Συρία, από τη μία πλευρά εμείς θα θέλαμε το καθεστώς να αλλάξει και ε, να αποσυρθεί, όπως πολύ σωστά το είπατε, και σας είμαι ευγνώμων για τις πρωτοβουλίες σας και τις πρωτοβουλίες του Αραβικού Συνδέσμου αλλά όσον αφορά τις μειονότητες και τις ε, χριστιανικές μειονότητες διαπιστώνω και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση της καταστάσεώς τους διότι υπάρχει μία εξέλιξη μίας επαναστατικής κινήσεως η οποία είδαμε και στην Αίγυπτο τι έγινε με τους κόπτες, τι γίνεται με το Σύνταγμα και ε, ενδεχομένως υπάρχει ακριβώς το αντίθετο, μία αρνητική εξέλιξη, αρνητικές επιπτώσεις και στις περιπτώσεις αυτές ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε λογικές εξελίξεις για τις ε, ανθρώπινες σχέσεις και προς όφελος αυτών οι οποίοι ζουν στην περιοχή. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, αρχίσω να απαντώ θα ήθελα να πω το εξής. Πώ αξιολογώ τον πρόεδρο της Συρίας. Όποιος έχει κάνει εγκλήματα ε, κατά ε, του λαού του θα πρέπει να ε, προσαχθεί στη διεθνή δικαιοσύνη. Κάποιος είπε προηγουμένως ότι έχουμε 17 συμφωνίες διμερείς και θα έχουμε και άλλες, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, είναι πολύ σημαντική. Και τα τελευταία 20 χρόνια το θέμα αυτό εκκρεμεί. Έχει έρθει η ώρα να έρθει σε αίσιο πέρας. Γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόρπου είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικό η συμφωνία αυτή να λιάνει το έδαφος για περισσότερες ε, σχέσεις εμπορικές ε, με τις χώρες της Ευρώπης. Τα σαλαφιστικά κινήματα και κατά πόσο είναι Ισλαμιστές και τρομοκράτες. Κοιτάξτε, οι σαλαφιστές δεν είναι τρομοκράτες. Εγώ δεν είμαι θεολόγος, αλλά είμαι περήφανος που είμαι μουσουλμάνος. Και ε, το σαλάφ ε, είναι κάτι ε, σαν καλή πράξη, μια καλή Ισλαμική πράξη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πιστοί, πιστεύουν στο Μωάμεθ, στον προφήτη και σίγουρα δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, ούτε κίνημα που επιζητεί τις δολοφονίες. Ε, αυτά αναμεγνύονται Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι θεολόγος, αλλά τα ζητήματα αυτά είναι ε, εύκολο να ε, οδηγήσουν σε σύγχυση. Και ξέρω ότι είναι και δημοφιλές να αναφέρουμε αυτά τα επιχειρήματα. Αυτά που σας λέω μπορεί να, να μην είναι αρεστά, αλλά δεν έχω έρθει για προεκλογική εκστρατεία Συγγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω ταυτόχρονα αραβικά και αγγλικά. Έχουμε τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Εάν ε, δεν μπορώ κάτι να εξηγήσω στα αραβικά, προσπαθώ να το εξηγήσω στα αγγλικά. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ε, ταυτίζουμε αυτόματα το Ισλάμ με την εγκληματική δραστηριότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί να γίνεται ε, ε, αυτή η περιττή σύγκρουση κάθε φορά. Ούτε είναι ηθελημένο. Πρόκειται για μικρές μειονότητες που χρησιμοποιούν ε, αυτές τις συγχύσεις που δημιουργούν προς ίδιον όφελος. Δηλαδή ταυτίζουν το Ισλάμ με την τρομοκρατία. Εδώ υπάρχουν καθεστώτα που επί 40 χρόνια δίωκαν τους Ισλαμιστές και τώρα έχουν φτάσει στην εξουσία αυτή λόγω της ανόητης και άσκοπης καταδίωξής τους και δίωξης. Σε όλες τις αραβικές χώρες υπάρχει το Ισλάμ και μειονότητες και είναι σημαντικό να προστατεύονται αυτές οι μειονότητες και σε καμία περίπτωση ε, δεν θα πρέπει να παραβιάζονται, να καταπιέζονται. Ούτε είναι γεγονός αυτό παντού είτε είναι χριστιανικές μειονότητε, είτε όχι. Ανήκουν στον κοινωνικό ιστό, ανήκουν στη χώρα, είτε είναι αυτή η Συρία είτε οποιαδήποτε άλλη αραβική χώρα. Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να ε, μην καταπιέζει ε, να καταπιέζει τις ε, μειονότητες. Σε ό,τι αφορά τις τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λιβύη που έχει μια ερώτηση σχετική. μετά από 42 χρόνια χάους λόγω του πρώην καθεστώτος δεν υπάρχει κανένα σύστημα, καμία τάξη, ε, κανένα κράτος στην Λιβύη. Έγινε επανάσταση και στη Λιβύη και στην Τινησία, αλλά δεν ε, επήλθε στην Τινησία το ίδιο χάος με τη Λιβύη, γιατί ε, στην Αίγυπτο και στην Τινησία υπάρχουν κρατικοί θεσμοί υπάρχει κράτος ε, που μπορούν να στηρίξουν αυτοί οι θεσμοί. Γι' αυτό η δομή και η διάρθρωση του κράτους δεν κατέρευσε. Στη Λιβύη δεν υπήρχαν θεσμοί. Υπήρχαν μόνο κάποιες ομάδες. Ούτε καν στο στρατό δεν υπάρχει ενότητα. Είναι πολιτοφυλακές, ομάδες κατακαιρματισμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν πρώτα απ' όλα οι Λίβοι για το πώς θα οικοδομήσουν το κράτος τους και τις κρατικές αρχές. Εκεί θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, όπως ε, έχουμε πράξει μέχρι τώρα. Ορισμένοι έχουν όφελος ε, και συμφέρον να χαρακτηρίζουν τους μεν Ισλαμιστές, μη Ισλαμιστές. Αυτό δεν ισχύει. Θα πρέπει να δούμε ποιος στηρεί τους κανόνες, ποιος στηρεί ε, τις ε, συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο και ποιος όχι. Όποιος δρά παράνομα θα πρέπει να αποτρέπεται από αυτή τη δράση. Είτε είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, ε, εβραίος κτλ. Όποιος δεν τηρεί το διεθνές δίκαιο δεν είναι σύμμαχός μας, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του. Ε, ε εμείς συνεργαζόμαστε με όποιον σέβεται και τηρεί τους νόμους, είτε είναι Ισλαμιστής, είτε είναι μουσουλμάνος. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι συνταγματική η δράση του και αν ανταποκρίνεται στην τάξη των πραγμάτων οι επαναστάσεις είναι γεγονός ότι ε, είναι δυναμικές καταστάσεις και μπορούν να κρατήσουν χρόνια. Ας πούμε, ε, η Πορτοκαλή επανάσταση και η επανάσταση του Twitter στην Αίγυπτο προήλθε από τη μεσαία τάξη και όχι από τα χαμηλά στρώματα ή από τους ανέργους. Από εκεί ξεκίνησε η επανάσταση. Γιατί ήταν τέτοιο το καθεστώς με κληρονομική κυβέρνηση. Υπάρχουν χώρες που είναι μοναρχίες και γνωρίζουν ότι έχουν ε, ε, βασιλιά. Κάποιος αναφέρθηκε στην Ιορδανία ή στο Μαρόκο και γνωρίζουμε τι ισχύει εκεί. Εγώ δεν είμαι υπέρ της μοναρχίας επειδή είμαστε μοιράτο, αλλά ε, οι μοναρχίες κατανοούν τον λαό γνωρίζουν το λαό, ε, ακούν τους πολίτες στο δρόμο. Ενώ ε, άλλες χώρες που είναι ε, δημοκρατίες ήθελαν να κληροδοτήσουν την κυβέρνηση, ας πούμε, στο γιο του Προέδρου. Με ρωτήσατε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Μας κατηγορούν ότι αναμειχθήκαμε και δώσαμε χρήματα στους σαλαφιστές και ποια ήταν και πόσα ήταν αυτά κτλ. Κοιτάξτε, εμεί δεν έχουμε κονδύλι στον προπολογισμό ούτε για σαλαφιστές, ούτε για κανέναν άλλον. Έχουμε ε, κοινοφελείς οργανώσεις στο Κατάρ, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές, που κάνουν εράνους στο λαό. Αλλά οι έρανοι αυτοί ελέγχονται πάρα πολύ από την Κεντρική Τράπεζα και από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας για να ε, πηγαίνουν, ας πούμε, στην οικοδόμηση ενός νοσοκομείου, ενός τεμένους, ε, στην ανέγερση ενός σχολείου, ενός χωριού κτλ. Βεβαίως δεν μπορώ εγώ σας εγγυηθώ 100% ότι δεν υπάρχουν καταχρήσεις ή παραβιάσεις. Γιατί και εσείς στις χώρες σας δεν έχετε κοινοφελή ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις που πηγαίνουν σε άλλους σκοπούς τα χρήματα που δεν θα δεγόσασταν εσείς ως ευρωβουλευτές ή ως ε, δημοκρατικές κοινωνίες. Καταχρήσεις υπάρχουν, αλλά εμείς φυσικά στη χώρα μας δεν έχουμε κονδύλι στον προπολογισμό για να υποστηρίσουμε ένα συγκεκριμένο κίνημα, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι Ε, ο κόσμος θα πρέπει να επιλέγει την κυβέρνησή του ελεύθερα. Και το Κοράνι λέει ότι κανείς δεν υποχρεώνεται σε, σε, τίποτα. Υπάρχει ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Ρωτήσατε και για την επέμβαση ε, στο Μπαχρέιν ε, των χωρών του Συμβουλίου του Περσικού Κόλπου τα στρατεύματα στο Μπαχρέιν δεν είναι του κατά. Υπάρχει μια παλιά συμφωνία ήδη από το 20, από το 30 μεταξύ ε, των χωρών για ε, στρατεύματα ταχείας επέμβασης για τη διαφύλαξη της ασφάλειας ε, των χωρών της περιοχής. Δηλαδή, αν μια χώρα χρειάζεται αυτά τα στρατεύματα, ε, ζητήσει τη βοήθεια και τη συνδρομή τους, θα πρέπει να αποσταλούν. Υπάρχει και νόμος μάλιστα που μας υποχρεώνει. Κάτι ανάλογο με το ΝΑΤΟ σε εσά για τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής. Ε, μας αναγκάζει ο νόμος να συνδράμουμε. Αλλά δεν είχαμε επέμβαση στρατιωτική. Πήγαν εκεί τα στρατεύματα για να προστατεύσουν κάποιες υποδομές στο Μπαχρέιν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο Μπαχρέιν. Υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε το παραδέχεται και η χώρα ίδια και προσπαθεί να το λύσει με τρόπο ειρηνικό και όσο γίνεται ταχύτερα. Διότι είναι ονίζεται αυτό το θέμα μεταξύ δύο ομάδων του λαού του Μπαχρέιν. Ο κύριος Μπασιούνι κατέθεσε μια διεθνή έκθεση. Γίνονται έρευνες για το ποιο παρενέβη τον νόμο, παραβίασε τον νόμο. Καλά, εγώ δεν θα μιλήσω εδώ εξ ονόματο του Μπαχρέιν, αλλά ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα στην περιοχή και οι έξωθεν ε, είναι ένα ζήτημα εκεί. είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να ε, φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των λαών με το διάλογο με ειρηνικό τρόπο και να ε, υλοποιούμε τις επιθυμίες τους. Γι' αυτού υψηλότης ο Εμμύρης του Κατάρ επαναλαμβάνει πάντα ότι οι μεταρρυθμίσεις είτε είναι άνωθεν είτε είναι κάτωθεν θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ειρηνικό και όχι με βομβαρδισμούς και με βιοπραγίες. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Δεν προσπαθώ ποτέ να αποφύγω τις ερωτήσεις, ακόμα και αν είναι δύσκολες ακαθόδεις. Εάν κάτι δεν απάντησα, σίγουρα δεν ήταν πρόθεσή μου. Α, για τις σκεφτικές μειονότητες στην Αίγυπτο. Ναι, ναι. Και την Παλαιστίνη. Κάτι με ρωτήσατε για την Παλαιστίνη. Όπως γνωρίζετε, το Παλαιστινιακό έχει έρθει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπάρχουν ε, ε, ψηφίσματα του Συμβουλίου ε, Ασφαλείας τα οποία δεν τηρεί το Ισραήλ. Εμείς θέλουμε ειρηνική επίλυση και δύο κράτη στα σύνορα του 1967. Η πολιτική του επικισμού θα πρέπει να τερματιστεί, διότι αν παραμείνει αυτή η σύγκρουση είναι η επόμενη ορολογιακή βόμβα, η επόμενη σπίθα που θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενναία. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ε, τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Και η, η γειτονιά του Ισραήλ έχει αλλάξει. Θα πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό το Ισραήλ. Οι αραβικοί λαοί και οι αραβικές κυβερνήσεις πλέον θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την κοινή γνώμη. Δεν μπορούν πλέον να την αγνοούν. Και αν συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, αυτή η διένεξη, είναι η επόμενη ορολογιακή βόμβα στην περιοχή. Γι' αυτό χρειάζεται ειρηνική επίλυση. Όχι όμως να επιβάλλει το Ισραήλ τη γνώμη του, αλλά βάσει του κράτους ε, δικαίου και του διεθνούς δικαίου τίποτα παραπάνω αλλά και τίποτα λιγότερο. Σας ευχαριστώ. إذا كان ممكن توقيع Ναι. Ε، κάτι άλλο που με ρωτήσατε είναι η συμφωνία για τους ανοιχτούς εθέρες, για τις εναέριες μεταφορές. Εγώ είμαι υπέρ ε, τέτοιων συμφωνιών είτε με την Ευρώπη είτε με τις ε, χώρες ε, του Περσικού κόλπου. Αυτό θα βοηθήσει, θα αυξήσει τον τουρισμό, τα ταξίδια, θα βοηθήσει για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των λαών Συμφωνώ, δεν μπορεί παρά να είναι θετική μια τέτοια συμφωνία και θα πρέπει να την προωθήσουμε. Και πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά θα τα διαβιβάσω στους συναδέλφους μου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, σας ευχαριστούμε που συζητήσετε μαζί μας με τρόπο τόσο ειλικρινή και ελπίζω να συνεχίσουμε αυτές τις σχέσεις και να παραμείνουμε σε επαφή διότι είμαστε ένα ο τμήμα του ίδιου κόσμου και μάλιστα στη γειτονιά μας έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα ε, και χαίρομαι για τη μελλοντική μας συνεργασία. Σας εύχομαι και πάλι καλή διαμονή στις Βρυξέλλες και καλή επιστροφή στην πατρίδα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.